Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αρχίζει καινούργια εβδομάδα. Η πρώτη τελευταία πριν τις πασχαλινές διακοπές. Κάτι που θα μας φτιάξει λίγο για τη διάθεση φαντάζομαι. Καλωσορίζω θερμότατα τους ευρωβουλευτές, τους ε, αγαπητούς καλεσμένους μας και όλους όσοι λαμβάνουν μέρος στη σημερινή μας συνεδρίαση. Στο πρώτο τμήμα της, ε, που είναι σήμερα το απόγευμα, θα συνεχιστεί όμως και αύριο πρωί και απόγευμα. Ως προς την ημερήσια διάταξη υπάρχουν μήπως παρατηρήσεις. Όχι. Οπότε να σας υπενθυμίσω ότι αναμεταδίδεται και από το διαδίκτυο η συνεδρίασή μα και έχουμε διερμηνία από και προ 20 γλώσσε με εξαίρεση τα εστονικά, μαλτέζικα, σλοβακικά και κελτικά γοδελικά. Περνάμε στο σημείο 3 της τη διάταξη που είναι το κυρίω θέμα τη απογευματινή μας συνεδρίας. Ένα εργαστήριο με θέμα τι συνέπειε των διαρθρωτικών αλλαγών στην Ευρωπαϊκή Γεωργία και πώς μπορούμε καλύτερα να στηρίξουμε το ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο στον 21ο αιώνα με την κοινή γεωργική πολιτική. Έχετε λάβει το πρόγραμμα αυτής της ακρόασης. Εξαιτία ε, του μεγάλου βαθμού διαστρωτική ποικιλομορφία τη ευρωπαϊκή γεωργία και οι δυναμικέ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ε, μπορούν να είναι πολύ διαφορετικέ το αναφέρουμε επανειλημμένως, γιατί αποτελεί και ένα βασικό πρόβλημα του ευρωπαϊκού γεωργικού μοντέλου. Είναι περίπλοκο φαινόμενο αυτών των διαφορετικών αλλαγών και έχει πολλούς παράγοντες που είναι αλληλένδετοι μεταξύ τους και επίσης διαφορετικούς κινητήριους μοχλούς. Θα πρέπει λοιπόν να, υιοθετήσουμε μια πιο περιεκτική γενικότερη θεωρία διαρθρωτικής ανάπτυξης τη γεωργίας. Και γι' αυτό η Επιτροπή μας μαζί με το Τμήμα Πολιτικών Β οργανώσαμε αυτό το εργαστήριο με θέμα τις συνέπειες των διαφορετικών αλλαγών στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Θα εξετάσουμε τις διάφορες ευρωπαϊκές πολιτικές επιλογές που προσφέρονται για στήριξη και καλύτερη ανάπτυξη του ευρωπαϊκού γεωργικού μοντέλου. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω εδώ και να ευχαριστήσω θερμά τους εκπροσώπους του Τμήματος Β, τμήματο Πολιτικών Β και την πολύ αγαστή συνεργασία που είχαμε σε ό,τι αφορά τη διοργάνωση αυτού του εργαστηρίου, αυτού του σεμιναρίου και για το πλούσιο υλικό που μας έδωσε και που μας επέτρεψε να εμβαθύνουμε και να αντριφήσουμε καλύτερα σε αυτό το περίπλοκο θέμα. Το σεμινάριο θα το διαιρέσουμε σε τρία τμήματα. Στο πρώτο τμήμα θα έχουμε τις διαφορετικές αλλαγές στη Δυτική Ευρώπη και την κοινή γεωργική πολιτική. Εδώ ο κύριος μας ομιλητής είναι ο κύριος ε, Γιάνν Ντόεβαντερ Πλούχ, που είναι ε, επικεφαλής της ε, έδρας της γεωργικής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Βάγκενιγκεν στις κατοχώρες. 20 λεπτά θα αφιερώσουμε στο τμήμα αυτό. Δεύτερο τμήμα αφορά τις διαφορετικές αλλαγές στη γεωργία στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη σε σχέση με την κυνηγιορική πολιτική. Περιφερειακή λοιπόν προσέγγιση οθετούμε όπως βλέπετε. Εδώ θα επικεντρωθούμε στις χώρες της μεγάλης διεύρυνση, στι 10 χώρες κεντρικής και Ανατολική Ευρώπης. Εδώ ο μιλητή μας είναι ο κύριος Ανικό Γιοχάς, που είναι ο Γενικό Διευθυντής του Ερευνητικού Ινστιτούτου Γεωργικής Οικονομίας από τη Βουδαπέστη. Και το τρίτο τμήμα του εργαστηρίου, του σεμιναρίου, είναι η επιστηστική αλυσίδα αξιών και πώς θα, βελτιώ, τη βελτιώσουμε και θα ενισχύσουμε τη διαπραγματευτική ισχύ των γεωργών. Εδώ ο μιλητής μας είναι ο κύριος Αλεσάνδρο Σορεντίνο, που είναι τακτικός καθηγητής ε, της γεωργοδιατροφικής οικονομίας από το Πανεπιστήμιο Τούσια της Ιταλίας. Έχουμε κορυφαίους εμπειρογνώμονες, πολύ αξιόλογους καλεσμένους και περιμένουμε τις ομιλίες τους που πιστεύω ότι θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις μας και θα μας επιτρέψουν να εξοικειωθούμε καλύτερα με το περίπλοκο αυτό φαινόμενο των διαρθρωτικών αλλαγών. Θα ακολουθήσουμε τη σειρά που σας παρουσίασα για τα διάφορα τμήματα του σεμιναρίου και σε αυτό το 20 λεπτό που διέθεσα στον καθένα παρακαλώ να παρουσιάσετε τις απόψεις και την ομιλία σας. Πρώτος έχει το λόγο ο καθηγητής από την Ολλανδία, από το Βάγκεν, είμαι ο κύριος Βαντεμπλούχ. Thank you very much, uh, Mr. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές. Με χαρά έρχομαι να συμμετάσχω στη συζήτηση αυτή για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Γεωργίας και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει και η γεωργική πολιτική σε αυτό. Έχω πέντε τμήματα ε, για την παρουσίασή μου. Πολύ σύντομα θα εξηγήσω ότι είναι οι διαρθρωτικές αλλαγές, ή εξελίξεις όπως τις λένε κάποιοι, μετά ποια είναι τα δεδομένα των τελευταίων δεκαετιών, τι στην πραγματικότητα συνέβη. Μετά θα στραφώ στην ε, ενίσχυση της σημασίας των μικρών μονάδων. Πολύ συχνά ξέρω ότι μιλούμε για αύξηση του μεγέθους των μικρότερων επιχειρήσεων, των μικρότερων μονάδων, αλλά ίσως δεν είναι ακριβώς τόσο περιορισμένη αυτή όσο μπορεί να φαίνεται. Δεύτερον, θα ήθελα να ανοίξω τη συζήτηση στο θέμα που ξεπερνάει, μάλλον σε μια θεώρηση που ξεπερνάει το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων, αλλά πάει προς στο τρόπο ε, άσκηση της γεωργίας, πώς γίνεται η οργάνωση, τα μέσα κτλ. Και εν τέλει με τα συμπεράσματα τι θα ήταν μια ανοιχτή ανάπτυξη της υπαίθρου. Καταρχάς λοιπόν διαστοτικές αλλαγές. Συνήθως σε τρία επίπεδα αναπτύσσουμε την έννοια των διαστοτικών αλλαγών. Η πρώτη αντίληψη είναι η ε, περιγραφική, τη γνωρίζουμε όλοι, εν προκειμένου πρόκειται για τον περιορισμό του αριθμού των ε, εκμεταλλεύσεων, μέσω μεγέθους των εκμεταλλεύσεων, όλο και πιο ε, λίγες μικρές εκμεταλλεύσεις και μεγάλες, μεγα, ε, πολύ, περισσότερες μεγάλες. Αυτό το έχουμε δει, ας πούμε, ξέρουμε ποια είναι η περιγραφική αντίληψη. Μετά υπάρχει μια οργανική αντίληψη, θεωρητική θα λέγαμε ίσως, η οποία υποθέτει βάσει της νέας κλασικής οικονομίας ότι μικρές επιχειρήσεις οι μικρές επιχειρήσεις είναι μικρές τόσο που δεν μπορούν να δώσουν απόδοση, επένδυση, ε, δυναμική στην οικονομία και ως εκ τούτου είναι καλύτερες ε, κερδοφόρες, ε, πρόσφορες επενδύσεις και τη βελτίωση της θέσης της η θέση επικεντρώνεται μόνο στη δραστηριότητα την επιχειρηματική, αλλά αυτό που λένε οι Γάλλοι, ε, γενική επιχειρηματική δραστηριότητα μιας ε, γεωργικής οικογένειας δεν λαμβάνεται υπόψη. Μόνο οι γεωργικές δραστηριότητες υπολογίζονται σε αυτή τη δεύτερη οργανική θεώρηση. Και τρίτον, ο στόχος, η γεωργική πολιτική με τους στόχους της διαθωτικής αλλαγής. Δηλαδή θεωρείται ότι είναι οι πόσες για το μέλλον οι μεγάλες επιχειρήσεις, ότι είναι οι μόνες οι οποίες μπορούν να ανθέξουν στον ανταγωνισμό της παγκόσμιας αγοράς, τις δύσκολες ε, συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς κτλ. Τρία επίπεδα λοιπόν για την, περιγραφή, για την ε, έννοια της διαθροτικής αλλαγής ή εξέλιξης. Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι αυτή η πρώτη η πρωτη έννοια είναι ορθή είδαμε στην περίοδο αυτή που ζούμε, στην εποχή μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή την εξέλιξη. Υπάρχουν και άλλες περίοδοι, ε, άλλες περίοδοι μπορεί να έχουν άλλες εξελίξεις κτλ. Αλλά αυτό που βλέπουμε στην Ευρώπη και τη Δυτική Ευρώπη θα μπορούσαμε να το συνοψίσουμε λέγοντας υπάρχει διαφορετική αλλαγή. Ε, ως προς την οργανική όμως αντίληψη, ότι δηλαδή είναι ε, απαραίτητο να εξαφανιστούν οι μικρές ε, εκμεταλλεύσεις και να ε, ενισχυθούν οι μεγάλες, εδώ μπορούμε να πούμε ότι είναι εσφαλμένη αυτή η, η αντίληψη. Είναι, είναι σφάλμα αντίληψης επίπεδου, όπως θα λέγανε οι επιστήμονες. Δηλαδή αυτό το οποίο μπορεί κανείς να διαπιστώνει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο δεν μπορεί να προβληθεί σε μονάδες παρατήρησης σε άλλο επίπεδο, μικρό επίπεδο ασφαλώς. Σε μάκρο επίπεδο μπορεί να βλέπουμε αύξηση μεγέθους εκμεταλλεύσεων και εξαφάνιση μικρών εκμεταλλεύσεων, χωρίς όμως αυτό απαραίτητα να συνεπάγεται ότι κάθε μικρή επιχείρηση, εκμετάλλευση θα εξαφανιστεί, ούτε ότι κάθε μεγάλη εκμετάλλευση θα ενισχυθεί. Δεν ισχύει δηλαδή σε κάθε επίπεδο αυτή η παρατήρηση. Και τρίτον, γιατί ο στόχο γεωργική πολιτικής, θέλω να σχολιάσω ότι η διαρθωτική αλλαγή βρίσκεται σε αντίφαση με τις ανάγκες της ε, κοινωνίας. Για να δούμε λοιπόν τα δεδομένα. Εδώ εστιάζουμε περισσότερο στι κάτω χώρε, αν και έχω και μια θεώρηση γενικότερη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εστιάζουμε στι κάτω χώρε καταρχά, γιατί πρόκειται για χώρα, όπω άλλωστε και η Δανία, όπου ε, ήταν ξεκάθαρη η διαρθρωτική αλλαγή. Και δεύτερον, διότι στι κάτω χώρε υπάρχει μια μοναδική βάση δεδομένων που επιτρέπει να παρακολουθήσουμε το ιστορικό των εκμεταλλεύσεων, μεμονωμένων εκμεταλλεύσεων, σε ε, μεγάλη ιστορική γραμμή. Και έτσι μπορούμε να έχουμε μια ε, ευρεία κλίμακα ανάλυσης. Συνήθως χρησιμοποιούμε δεδομένα από αλλά εδώ έχουμε άλλη βάση δεδομένων που μας επιτρέπει και διαφορετικές αναλύσεις. Και Φερρυπίν θα κοιτάξω ε, σε μια μικρή επιχείρηση που μπορεί να αναπτυχθεί αν δουλεύει ο γεωργός σκληρά, να γίνει μεσαίου μεγέθους και αργότερα και μεγάλου μεγέθους και έτσι από τη μία στη δεύτερη απογραφή να εξαφανιστεί. Εξαφανίζεται από τι στατιστικέ. Δεν είναι μικρή επιχείρηση. Δεν είναι μικρή εκμετάλλευση. Γιατί, γιατί έγινε μεσαία εκμετάλλευση, με ξέρω μεγέθου και μετά έγινε μεγάλου μεγέθου. Άρα αυτού του τύπου οι ε, απογραφέ δεν μπορούν να καταγράψουν τι δυναμικέ των στατιστικών. στη δική μου τη στατιστική, στατιστικά μου τα δεδομένα, το, μπορώ να το παρακολουθήσω αυτό από το 80 έως το 2006 είναι τα δεδομένα, αφορούν ε, βοσκοτόπια και αρρώσιμες εκμεταλλεύσεις, ε, ζώα βοσκής. Έχουμε δεδομένα καθαρού μου επιδότησης, άρα σε, μέγεθους, σε μονάδες μέγεθους ε, κάτω χωρών και καταγραφεί τόσο το σημείο κίνησης, κατάσταση εκκίνησης, όσο και η εξέλιξη στον χρόνο. Είναι πιο εύκολο να μεταβούμε στην επόμενη διαφάνεια που δείχνει ποια είναι, ποια είναι η δυναμική του χρόνου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κοιτάξουμε στην πρώτη, που έχουμε 10 με 50 ε, καθαρά ισοδύναμα επιδότησης, στην περίοδο 80-90, μικρές επιχειρήσεις λοιπόν, μικρές εκμεταλλεύσεις, μετά έχουμε τις μεσαίου μεγέθους, τις μεγάλες τρεις διαφορετικές ε, κατηγορίες μεγέθους, μικρές, μεσές, μεγάλες εκμεταλλεύσεις, ανάλογα με, τις, τον αριθμό των αγελάδων και στην περίοδο αυτή έχουμε αυξήσεις σε μέγεθος των μικρών ε, εκμεταλλεύσεων αλλά και μειώσεις. Το ίδιο μάλιστα και για τις μεσαίου αλλά και για τις μεγάλου μεγέθους. Έχουμε μερικές που μίκριναν συρρυκνώθηκαν. Επίσης έχουμε την εσωτερική, την κυκλική ροή εξέλιξη των ε, εκμεταλλεύσεων, μικροσκοπικές που μπαίνουν μετά στην ε, μικρού μεγέθους ε, και πέραν του outflow της εξωτερικής ροής υπάρχει και η εσωτερική ροή και ισχύει για όλα τα μεγέθη αυτό, όπως και η διαρροή από τις μικρές στις μεσαίου μεγέθους εκμεταλλεύσεις, οι 10 έως 50 μονάδες γίνονται 5 έως 100 και μετά μπορεί ακόμη και να προχωρήσουν στην κατηγορία του μεγάλου μεγέθους. Υπάρχουν και πολλαπλές δυναμικές, μπορεί μικρές εκμεταλλεύσεις να εξαφανιστούν, εξαφανίζονται όμως και μεγάλες επιχειρήσεις, όπως και μπορούν μεγάλες επιχειρήσεις να αυξηθούν, να ενισχυθούν, όπως μπορούν να ενισχυθούν και μικρές εκμεταλλεύσεις. Αυτό σημαίνει πολλαπλή δυναμική. Και επίσης, και σε αυτό καταλήγω σε ένα πολύ ενδιαφέρον ε, συμπέρασμα, ότι η μικρή εκμετάλλευση της τωρινής εποχής μπορεί να είναι μεγάλη εκμετάλλευση στο μέλλον. Δεν αποκλείεται δηλαδή μικρές εκμεταλλεύσεις να εξελιχθούν περαιτέρω, μπορούν να αλλάξουν κατηγορία, να γίνουν μεσαίου μεγέθους και ακόμη και μεγάλες. διότι θα έχουν εξαφανιστεί περισσότερες μεγάλες επιχείρησεις και ελάχιστη κατηγοριοποίηση. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της δυναμικής. Και επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η δυτή ε, εξέλιξη. Εδώ βλέπετε στο πρώτο κομμάτι την ενίσχυση του μεγέθους των μεγάλων εκμεταλλεύσεων και τις ε, μικρές που μικραίνουν ακόμη περισσότερο. Αυτή είναι η παραδοσιακή, η συμβατική καλύτερα θεώρηση, ενώ η εμπειρική θεώρηση είναι ότι υπάρχουν διπλές τάσεις, διτές τάσεις και στις δύο κατηγορίες. Βέβαια υπάρχουν ε, διαφορετικές ε, λογικές από αυτό. Η μία είναι η οικονομική λογική και η άλλη είναι η κοινωνική ε, λογική. Δηλαδή η οικονομική λογική μπορεί να λέει ότι ενισχύεται, αναπτύσσεται η εκμετάλλευση, αλλά μπορεί και για λόγους οικονομικών δυσχεριών να εξαφαλιστεί κάποια στιγμή, κάτι το οποίο θα σας δείξω αργότερα. Είναι η κοινωνική λογική λέει ότι ο, ο νέος Γεωργός αφοσιώνεται στην ε, εκμετάλλευσή του, θέλει να τη μεγαλώσει, θέλει να παραμείνει αυτόνομη κτλ. Και αναπτύσσει εκ τούτου την εκμετάλλευση. Ταυτόχρονα η κοινωνική θεώρηση μπορεί να οδηγήσει και στην αντίστροφη, στο αντίστροφο συμπέρασμα. Δηλαδή ότι κανεί αρχίζει και απογοητεύεται, βλέπει ότι η δουλειά αυτή είναι πολύ μονότονη και τελικά καταλείπει την ε, εκμετάλλευση. Όλα αυτά για να πω ότι είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς εκ των προτέρων τι μπορεί να ε, συμβεί. Εδώ το μόνο που μπορούμε να δείξουμε ότι υπάρχει μία τάση εν γέννη να ε, αυξάνεται το μέγεθο των, των εκμεταλλεύσεων, υπάρχει ένα ανώτερο και ένα κατώτατο επίπεδο. Φαίνεται λίγο πολύ σαν να κάνουν βήματα χορού στο χρόνο μέσα οι εκμεταλλεύσεις, ενώ άλλε μειώνουν το μέγεθός τους, κάποιες άλλε μπορεί να μεγαλώνουν, κάποιες άλλε μπορεί και να εξαφανίζονται, κάποιε μπορεί να είναι ε, νέο εισερχόμενοι στην αγορά. Είναι πολλαπλή δυναμική δηλαδή. Δεν είναι μονογραμμική η εικόνα. Βεβαίως θα μου πείτε, α ναι καλά μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές, διαφορετικές ε, ανά πάσα στιγμή εξελίξεις και οι μεγάλες επιχειρήσεις να μεγαλώσουν και οι μεσές και οι μικρές και όλες ανά πάσα στιγμή μπορεί να ε, εξαφανιστούν. Εν πάση περιπτώσει τι σημασία μπορεί να έχει όλο αυτό. Να σας πω, εδώ έχουμε ακριβώς τα δεδομένα που δείχνουν από το 1980 στο 2006 την περίοδο περίπου 2,5 δεκαετιών τι συμβολή στη συνολική γεωργική ανάπτυξη στις κάτω χώρες των διαφορετικών ομάδων μεγέθους. Μικρές λοιπόν και μικρότερες από 50 μονάδες, ε, μεσές, πολύ μεγάλες και υπερμεγέθης εκμεταλλεύσεις. Οι μικρές λοιπόν συμβάλλουν κατά τετραπλάσιο στην συνολική γεωργική ανάπτυξη του γεωργικού τομέα στις κάτω χώρες από ότι οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις. Αυτό σημαίνει, όπως είπα, στο γεωργικό τομέα στις κάτω χώρες, αλλά ασφαλώς ισχύει και σε άλλες γεωργικούς τομείς, είναι σαν να μην βλέπουμε τον, ε, την ε, πραγματική δύναμη και κρυφή ενδεχομένω μυστική δύναμη του γεωργικού τομέα κατά χώρο, ότι δηλαδή έγκυται στι μικρέ και μεσαίου μεγέθου εκμεταλλεύσει. Και άρα πάμε στο διπλό παράδοξο τη ιστορική καμπή, που πάλι πλήττεται από αυτό το παράδοξο, ότι δηλαδή οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις οι οποίες καταρχήν είναι αυτέ που θα πρέπει να δείξουν ανταγωνιστικότητα ή θεωρείται ότι θα είναι σε θέση να αναπτυχθούν ε, αυτόνομα κτλ. Είναι αυτές οι οποίες τραβούν το πιο πολύ χρήμα. Πρώτο παράδοξο. Και δεύτερο, δεύτερο μέρος του παραδόξου, οι μεγάλες αυτές εκμεταλλεύσεις συμβάλλουν σχετικά λίγο στην συνολική ανάπτυξη και τη συνολική δυναμική. Πολύ παράδοξο το διπλό αυτό παράδοξο, και όταν λέμε ότι χρειάζεται περισσότερη ανάπτυξη, απασχόληση, εισόδημα που θα παράγουν οι εκμεταλλεύσεις, είναι προφανές ότι πρέπει με την προσεχή γενιά αυτής της ιστορικής καμπής να ξεπεράσουμε το διπλό παράδοξο. Και τώρα από το μέγεθος περνάω στο ύφος ε, της εκμετάλλευσης, ε, της γεωργικής δραστηριότητας. Έχουν γίνει έρευνες στην Ιταλία, την Ισπανία, την ε, Ιρλανδία, τις κάτω χώρες στην Αυστρία, που δίνουν διαφορετικά Ήθη γεωργικής εκμετάλλευσης και παραγωγής, είτε μπορεί κανείς να επιδιώξει την υψηλή τεχνολογία, είτε την παραδοσιακή μέθοδο, μεγάλη κλίμακα, περιορισμένη κλίμακα. Σε μακροπρόθεσμη λοιπόν έρευνα, όπως είναι τα στοιχεία που μας δίνουν οι κατοχώρες, βλέπουμε ότι και πάλι σε μια ε, πειραματική σύγκριση μεταξύ διαφόρων ε, υφών ε, γεωργικής εκμετάλλευσης με χαμηλό κόστος και high-tech, υψηλής τεχνολογίας δηλαδή, που συγκρίνονται μεταξύ τους ε, σε περίοδο δεκαετίας με, δύο, με βάση δύο διαφορετικά και αρχές σχεδιασμού δηλαδή πρέπει να έχει έναν γεωργό υπεύθυνο, δηλαδή ένας μόνο να κάνει όλη τη δουλειά και παραγωγή του ίδιου εισοδήματο από, την από την κάθε εκμετάλλευση. Αλλά το ίδιο εισόδημα με έναν μόνο ε, που δουλεύει την, επιχείρηση την εκμετάλλευση θα πρέπει να γίνεται είτε με χαμηλό κόστο, είτε με υψηλή τεχνολογία. 400.000 λοιπόν κιλά γάλακτο σε παραγωγή ορίστηκε ως επίπεδο ε, για την εξασφάλιση ενός αποδεκτού εισοδήματος για τις ε, εκμεταλλεύσεις χαμηλού κόστους, ενώ 783.000 φαίνονταν να απαιτούνται για μια ε, εκμετάλλευση ψηλής τεχνολογίας για να παραχθεί το ίδιο εισόδημα. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι στη, το εισόδημα από την εργασία για την παραγωγή των 400.000 ήταν μεγαλύτερο από το κόστος και αντίστροφα στην υψηλή τεχνολογία ήταν μικρότερο το ε, εισόδημα από την εργασία, αλλά το τελικό αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Εδώ τώρα βλέπουμε σε σχέση με τις τιμές. Μια πτητικότητα έχουν φτάσει μέχρι το 24. Η εκμεταλλεύσεις χαμηλού κόστους φαίνεται να κρατούν ένα επίπεδο, ενώ οι υψηλές τεχνολογίες έχουν αρνητική πλέον ρευστότητα. Ε, μέχρι το 2008-2009 βλέπουμε αυτή την κατάσταση με μια εξέλιξη αυτή τη στιγμή προς το αρνητικό. Κατάσταση παρατηρείται και στις κατοχώρες αλλά και στη Δανία με σημαντικό ποσοστό εκμετάλλευση των μεγάλων εκμεταλλεύσεων ή κλεισίματος. Γιατί στη νέα αυτή περίοδο των παγκοσμιοποιημένων και απορρεπτημισμένων ε, αγορών η πάλι πολύ ισχυρή και μεγάλη εκμετάλλευση φαίνεται πια μικρή και έχει υψηλό κόστος οικονομικό και δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την πτυτικότητα της αγοράς ενώ η μικρότερη εκμετάλλευση είναι σε θέση περισσότερο να ανθέξει αυτή την ε, πίεση. Στο, στα συμπεράσματα τώρα, παρά τις δεκαετίες επιλεκτικών γεωργικών πολιτικών, μικρές και μεσές εκμεταλλεύσεις παραμένουν ε, και επίσης αποτελούν προπύργια διαφύλαξης της ασφάλειας της επιστηστικής της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην νέα αυτή περίοδο αυτών των απορριθμισμένων αγορών οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις υψηλής τεχνολογίας, τεχνολογίας εχνής, είναι πιο ευάλωτες, είναι δηλαδή ο αδύναμος κρίκος στην ε, εξίσωση. Ενώ οι μικρές και μεσές επιχειρήσεις, επειδή είναι πιο πολυλειτουργικές, επειδή, πολυλειτουργικές, επειδή είναι ενσωματωμένες σε, μια ευρύτερη, σε ένα ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων, είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα την θετικότητα και εν τέλει αυτή η προτίμηση της προηγούμενης ε, κουγουπού για τις μεγάλες ε, επιχειρήσεις, ε, για τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις φαίνεται να είναι αναχρονιστική πλέον. Οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις όντως τώρα δυσκολεύονται να σεβαστούν τις ανάγκες για την ποικιλία, για την προσία του τοπίου, για την, την προσαρμογή στη νέα πολιτική, για την προστασία της υπαίθρου, την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών προσαρμογή στη χρήση του πόσιμου νερού ή του μη θαλασσινού νερού, την εξοικονόμηση ενέργειας, την ακόμα και την παραγωγή απασχόλησης, ακόμα και, παράδοξο αυτό πάλι, φαίνεται να μένει σε θέση να γίνονται πιο καινοτόμε από ότι οι μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις. Και το, τώρα για να περιγράψουμε σε ένα νέο πλαίσιο ε, πολιτικής αυτά τα ευρήματα, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πολύ απλά ότι αντί να είναι επιλεκτική η προσεχή που θα πρέπει να είναι ανοιχτή, περιεκτική, να δίνει δυνατότητες για κάθε ε, τύπο και μέγεθος εκμετάλλευσης, γιατί αυτή η διακριτική επιλογή, η διακριτική πτυχή δεν αντιστοιχεί στις ε, υφιστάμενες τώρα ανάγκες. Χρειάζονται βεβαίως κίνητρα για τις εκμεταλλεύσεις χαμηλού κόστος, όπως έδειξε η απόπειρα της Γαλλίας να πάει προς μια οικονομία ε, γεωργικών, οικολογικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και ε, να δοθεί ένα περιθώριο ανάπτυξης μικρών και με, των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, αλλά και ταυτόχρονα η καταποκοπή ενισχύσεις να συνδεθούν με την προστασία του τοπίου και της βιοποικιλότητας. Η ασφάλεια για την ε, παραγωγή των τροφίμων σημαίνει ταυτόχρονα ότι πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη πιστρών αγορών. Χρειάζεται υποστήριξη της ροής, της εισροής στο επάγγελμα νέων ανθρώπων και συμβολή στην αναδιατύπωση ενός θεματολογίου με στόχους για την κοινή γεωργική ε, έρευνα και ανάπτυξη. Και Πρόεδρε, ελπίζω να μην σας καθυστέρησα πολύ. Ευχαριστώ πολύ την προσοχή σα. Περνάμε στην επόμενη καλεσμένη μας. Νομίζω ότι τα χειροκροτήματα ήταν ο καλύτερος τρόπος ε, της επιδοκιμασίας και του θαυμασμού για την παρουσίασή σας. Περνάμε στην ε, κυρία Γιούχας την δεύτερη μας ε, εμπειρογνώμονα από την Ουγγαρία. Σας ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι. Έχω 15 ετή και εμπειρία ως επιστήμον και καθ' όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου έκανα ομιλίες ε, σε πολλά, πολύ μορφό κοινό, σε σε γεωργούς που ήταν το πιο δύσκολο κοινό, σε φοιτητέ, το ίδιο, σε υπαλλήλους, αλλά πρώτη φορά μιλώ σε πολιτικούς και παρακαλώ σας θέλω παρακαλώ να δείξετε υπομονή. Και μετά θα σας βαθμολογήσω όλα για να δω προς τη δυσκολία τι κοινό ήσασταν. Εγώ θα σας μιλήσω για τις διαρθρωτικές αλλαγές περισσότερο στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αυτές που παρατηρήσαμε την τελευταία δεκαετία. Και αυτή είναι η δομή της ομιλίας μου, της παρουσίας που θα σας κάνω. Πρώτο σημείο, ο στόχος της έρευνας. Ο στόχος της έρευνας είναι να κάνει μια περιγραφική αλλαγή των αλλαγών στις ε, διαρθρώσεις των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και να εξηγήσει τις κινητήρες δυνάμεις αυτών των αλλαγών, ε, καθώς και να αξιολογήσει κάποια, κάποιες άγουσες ανάπτυξης στις χώρες αυτές και να ε, σκεγγραφείς και κάποιες μελλοντικές πολιτικές για να προωθήσει μια πιο ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη. Καταρχήν ε, δώσαμε μάχη ε, ως προς τα δεδομένα. Χρειάστηκε να πασχίσουμε για να συνδυάσουμε τα δεδομένα από τη Eurostat, ιδιαίτερα την έρευνα για τις γεωργικές διαρθρώσεις, τους οικονομικούς οργανισμούς γεωργίας και το δίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης. Αυτές είναι οι βασικές βάση δεδομένων που γνωρίζουμε και είμαστε ιδιαίτερα εξοικειωμένοι στο Ερευνητικό μου Ινστιτούτο. Προσπαθούμε όμως να κάνουμε μια συνεκτική, συγκριτική ανάλυση μεταξύ των χωρών της Κεντρικής και Ανατολική Ευρώπης με τις ε, βάσει αυτές των δεδομένων. Παρόλο που πασχίσαμε, άλλοι συνάδελφοι καταρακώθηκαν και δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν καλά αυτές τις βάσει δεδομένων. Βέβαια θα πρέπει να αναπτύξουμε καλύτερα τα στατιστικά μας συστήματα για να τα κάνουμε πιο συνεκτικά και πιο επίκαιρα ως προς την ισορροή των πληροφοριών για να γίνει ε, δυνατή και συγκριτική ανάλυση μεταξύ των διαφόρων χωρών. Αυτό ήταν το έργο της ε, έρευνας, να μιλήσουμε για μικρές, μεσαίες και μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Ο περιορισμός των δεδομένων οφειλόταν στο γεγονός ότι στην ε, περίοδο που διερευνήσαμε είχαμε σημαντικές αλλαγές των στατιστικών στοιχείων σε μερικές χώρες τα φυσικά κατόφλια ήταν αποκλειστικά και δεν ήταν σταθερά σε μερικές χώρες. Πολωνία, Τσεχία και Σλοβακία για παράδειγμα. Στην Βουλγαρία περιληφθήκαν και τα βοσκοτόπια, οι λιμόνε το 2010 και αυτό μα δυσκόλεψε. Επίσης ε, η διαφορά μεταξύ του φυσικού μεγέθους ε, σε σχέση με το, τη μέση απόδοση είχε σημαντικές διακοιμάνσεις, κάτι που δημιούργησε πρόβλημα με τα δεδομένα του δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης. Επίσης είδαμε ότι αν διαλέξουμε δείκτες από τα δεδομένα αυτά, τα δεδομένα τα ίδια επηρεάζουν τα αποτελέσματα. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε τα συστήματα δεδομένων μας για να επιτρέψουμε καλύτερες αναλύσεις για τις διαρθρωτικές αλλαγές. Πάντως βλέπουμε γενικώ και κατά μέσο όρο ότι οι γεωργικές εκμεταλλεύσει και στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αυξάνουν σε μέγεθο, μειώνουν σε αριθμό και γίνονται πιο ε, μεγαλύτερη ένταση κεφαλαίου. Αυτό το βλέπουμε και στη Δυτική και στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Περισσότερε είναι πάνω από το μέσο όρο, πολλέ είναι στο μέσο όρο και οι λίγες είναι στο μεγάλο. Έχουμε λίγες λοιπόν μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε ό,τι αφορά την παραγωγή και έχουμε μεγάλο αριθμό μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Επίσης, ε, λίγε είναι οι μεσαίου μεγέθου γεωργικές εκμεταλλεύσει, οπότε δεν υπάρχει ουσιαστικά. Είναι, δύσκολο να βρεθεί ο μέσο όρο. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει, αλλά είναι δυσέβρετο. Και στι αναλύσει συνήθω μιλούμε για μέσους όρου. Πάντως ήταν πολύ καλή η προηγούμενη ομιλία που έδειξε την κοινωνιολογική άποψη μεταξύ των δύο διαφορετικών ομάδων, των μικρών και των μεγάλων. Πάντω, ε, λίγες ε, ήταν οι μεγάλες και έντες κεφαλαίου γεωργικέ εκμεταλλεύσει στην κεντρική στην και ανατολική Ευρώπη. Και εδώ βλέπετε τα στοιχεία. Η γαλάτια στήλη είναι αυτή της Ανατολικής Ευρώπης, των 10 χωρών της μεγάλης διεύρυνσης, με εξαίρεση την Κροατία, γιατί παραδίκαια αργά και δεν μπορέσαμε να τις περιλάβουμε στα στρατηγικά στοιχεία και η Μάλτα και η Κύπρος ε, δεν εμπίπτουν στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Βλέπετε πάντως γενικώ ότι μειώθηκε ο ρυθμός των ε, ε, γεωργικών εκμεταλλεύσεων και το μέσο μέγεθος αυξήθηκε, το μεσαίο μέγεθος των εκμεταλλεύσεων. Επίσης, μεγαλύτερη μείωση του εργατικού δυναμικού. Και αν δείτε τις, α, ε, τις γκρίζες, ε, τους γκρίζους βλέπετε ότι οι τάσεις ήταν βέβαια ταχύτερες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, αλλά απέχουμε ακόμη πολύ από την ε, Ανατολική Ευρώπη. Είχαμε 7,8 σε σχέση με το 8,1, οπότε έχουμε ακόμη κάποιο δρόμο να διανύσουμε. Επίσης, στις γαλάζιες στήλες που δείχνουν τις χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, βλέπετε ότι έχουμε τρεις μεγάλες γαλάζιες στήλες. Δύο από αυτές είναι στα αριστερά μου, για σας είναι στα δεξιά Εκεί έχουμε τη μείωση. Τι μειώνεται λοιπόν. Ο αριθμός των μεικτών καλλιεργειών και των ε, ε, εκμεταλλεύσεων που έχουν κτηνοτροφία και των μεικτών με καλλιέργειες και κτηνοτροφία, με γεωργία και κτηνοτροφία. Αυτό είναι που μειώνεται. Τι αυξάνεται. Αυξάνεται η τελευταία γαλάζια γραμμή στο κάτω μέλος που είναι οι υπαίθρες καλλιέργειες, οι αρρώσιμες καλλιέργειες που είναι ελαιούχες και πρωτεϊνούχες καλλιέργειες κυρίως. Αυτή είναι η μέση όρη λοιπόν. Και οι περισσότερες από τις θέσεις αυτές οφείλονται στην κοινή γεωργική πολιτική. Και εδώ βλέπετε τι συνέβη. Τώρα, γιατί, ποια είναι τα αίτια, ποιε είναι οι κινητήριε δυνάμει αυτών των αλλαγών. Αναφέρθηκα πρώτα στην κοινή γεωργική πολιτική. Έχουμε και την ε, παραγωγικότητα, το κοινωνικό πλαίσιο της ε, εκτός της ε, γεωργικής εκμετάλλευσης, ευκαιρίες απασχόλησης, χρήση γης, αγορά, μακροοικονομικό πλαίσιο, συλλογικές δράσεις και ούτω καθεξή Όλα αυτοί οι παράγοντες επηρέασαν τις αλλαγές στις διαρθρώσεις της γεωργικές. Επίση, αυξήθηκε η παραγωγικότητα στις χώρες της μεγάλης κυρίω ε, κυρίως εξαιτία τη ΚΑΠ και άλλων διαστρατικών αλλαγών. Αν δούμε όμω τη μέση απόδοση, βλέπουμε ότι στερεί σε σχέση με τις παλιές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15. Πάντω λίγε είναι, επαναλαμβάνω, οι ιδιωτικέ εκμεταλλεύσει ε, που βρίσκονται στο μέσο όρο. Και οι μεγάλε ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι υψηλέ τεχνολογίας γεωργικές εκμεταλλεύσει στην Ουγγαρία μοιάζουν αυτέ τι. Ολλανδία. Οι υπόλοιπε όμω είναι πολύ κάτω από το μέσο όρο. Επίσης αυξήθηκε και η ανταγωνιστικότητα. Τώρα εξάγουμε κυρίως ε, ε, βασικά αγαθά και πρωτογενό και δευτερογενό μεταποιημένα προϊόντα. Οι αγορέ μα έχουν γίνει πιο ε, ανταγωνιστικέ, αλλά εξακολουθεί να παραμένει μια διαφορά, ένα χάσμα που θα πρέπει να το καλύψουμε, να το γεφυρώσουμε για να βελτιωθούμε περαιτέρω. Επίση, βελτιώθηκαν τα γεωργικά εισοδήματα. Υπήρξε μια τέτοια βελτίωση. Και υπάρχει και μεγαλύτερη ανάπτυξη, ταχύτερη από τις, τις χώρες, 15 χώρες αρχικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά παρόλα αυτά υστερούμε. Και η βελτίωση οφείλεται κυρίως στις αρρώσιμες καλλιέργειες, δηλαδή στη γη, στην εκμετάλλευση της γης και στην παραγωγή των δημητριακών κυρίως σε μια συνάντηση γεωργών σε ένα εργαστήριο πριν μπω καν στην αίθουσα, στο κτίριο που γίνεται αυτή. βλέποντα μόνο το πάρκινγκ, το χώρο στάθμευσης, ε, καταλαβαίνω ποιο λαμβάνει μέρο σε αυτή τη συνεδρίαση. Αν όλα τα αυτοκίνητα στο πάρκινγκ είναι μεγαλύτερα και καλύτερα από το δικό μου, κάτι που συνήθω ισχύει, οι περισσότεροι είναι ε, καλλιεργητέ με αρρώσιμε καλλιέργειε, με υπαίθριε. Όταν έχουμε και χειρότερα και καλύτερα ε, αυτοκίνητα σημαίνει ότι δεν έχουμε μόνο γεωργούς, αλλά έχουμε και κτηνοτρόφους, κτηνοτρόφους, λησοκόμους Πάντως, ε, έτσι καταλαβαίνουμε τη σύνθεση αυτών των συνεδριάσεων, των συναντήσεων γεωργών. Επίσης, υπάρχει μια δημογραφική γύραση, κάτι που δεν είναι το ίδιο με τη Δυτική Ευρώπη. Γιατί στι αρχέ τη δεκαετία του 90, από αρχέ δεκαετία του 90 έχουν περάσει 25 χρόνια. Στι αρχέ τη δεκαετία του 90, στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ποιος απέκτησε μεγαλύτερη σημασία ή το εργατικό δυναμικό που ήταν γύρω στα 30 με 40 έτη. Τώρα αυτοί πηγαίνουν στη σύνταξη και δεν έχουμε οικογενειακές παραδόσεις μεταβίβαση της κοιτάλης από τη μία γενιά στην άλλη. Δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει ανανέωση. Γι' αυτό έχουμε και μεγαλύτερο πρόβλημα γύρασης του γεωργικού πληθυσμού στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Έχουμε πολλούς, έχω πολλούς συνομήλικους που θα μπορούσαν να πάρουν τη σκητάλη, αλλά είναι δύσκολο αν δεν έχουν ε, οικογενειακή εκμετάλλευση, αν δεν υπάρχει οικογενειακή παράδοση. Είναι πολύ δύσκολο ε, για τους ε, νέους γεωργούς να βρουν τέτοιες καλλιέργειες για να αναλάβουν και για τους παλιούς να μεταδώσουν, να μεταβιβάσουν την κληρονομιά. Επίσης, οι επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο δεν έτυχε ιδιαίτερη προσοχής στην προηγούμενη περίοδο και βλέπουμε τα αποτελέσματα, τα αρνητικά αποτελέσματα τώρα στο ότι δεν είχαμε επενδύσει σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Έχουμε ανειδίκευτου ε, στη Γεωργία δυστυχώς πολλούς, όχι ιδιαίτερα μορφωμένου. Ε, δεν υπάρχει συνεργασία, μεγάλος κατακαιρματισμός. Ε, δεν έχουμε πολλές ε, νομότυπες ε, εμπορικές δραστηριότητες. Έλλειψη χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου και αμοιβέ εμπιστοσύνη επίσης ε, εμποδίζουν τη συνεργασία. Και εδώ δεν μιλούμε για την έλλειψη εμπιστοσύνη στην κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά την πτώση του τείχους. Έχουμε ένα νέο είδος δυσπιστίας. Δεν είναι η παλιά δυσπιστία για τα κολχός. Επειδή οι παλιές ε, οργανώσεις και συνεταιρισμοί απέτυχαν, οι νέοι συνεταιρισμοί επίσης ε, αποτυχάνουν λόγω της δυσπιστίας που σώβει. Δύσκολη λοιπόν η συνεργασία. Ε, μερικές κινητήρες δυνάμεις ε, επιταχύνουν τις διαρθρωτικές αλλαγές και άλλα αίτια τις επιβραδύνουν. Αυτό δεν είναι τίποτα καινούργιο ή τίποτα παράδοξο ή εντυπωσιακό. Τι προτείνουμε όμως. Για τις άμεσες ενισχύσεις έχουμε δύο είδη. Έχουμε τα αποτελέσματα των άμεσων επενδύσεων που είχαν θετικό αντίκτυπο στα γεωργικά εισοδήματα, όπως σας είπα και προηγουμένως. Έχουμε όμως ε, μία αρνητική συνέπεια στην ένταση του εργατικού δυναμικού. Για μας, για την κυβέρνηση και τους επιστήμονες δεν είναι και πολύ αρνητική αυτή η τάση, γιατί σημαίνει ότι μπορούμε να κρατήσουμε την απασχόληση στην ύπεθρο σε υψηλότερο επίπεδο από ό,τι με άλλους τρόπους. Επίσης, οι συνέπειες δεν είναι ομοιόμορφες ε, στις επιχειρήσεις και στις περιφέρειες. Έχουμε διαφορετικά παραδείγματα στην Πολωνία, Σλοβακία, Ρουμανία, Τσεχία και υπάρχουν διαφορές ε, στην, ε, στις πληρωμές κατά μονάδα και στο φυσικό μέγεθος και στη γεωγραφική τοποθεσία. Πάντως γενικώ, οι άμεσες επενδύσεις στα μέσα της αγοράς και οι διεθνείς εξέλιξεις αγορές οδήγησαν σε αλλαγές στις διαρθρώσεις της παραγωγής κυρίως στις ανταγωνιστικές ε, αρρώσιμες καλλιέργειες που γίνονται και πιο δημοφιλείς. Επίσης, η πολλαπλή συμμόρφωση και το πρασίνισμα της ΚΑΠ δεν είναι βασικές κινητήρες δυνάμεις, ακόμη τουλάχιστον των διαρθρωτικών αλλαγών. Το 2015 ήταν η πρώτη χρονιά του πρασινίσματος και βλέπουμε περίπου 20% των Γεωργών να μπερδεύουν ε, τη, τις ανάγκες του πρασινίσματος ε, και των ε, περιοχών οικολογικής εστίασης και το χαρακτηρισμό τους. Πιστεύουμε ότι αργότερα θα εξοικειωθούν οι γεωργοί με το νέο σύστημα και θα βελτιωθούν μακροπρόθεσμα. Παρά τα λάθη που διαπιστώνουμε τώρα. Τώρα, ανάπτυξη της υπαίθρου και πώς τη στηρίζουμε στις 10 χώρες μεγάλης διαβρύσης. Έχουμε κάποια επενδυτικά προγράμματα για την αύξηση της παραγωγικότητας και την επίσπευση των διαστρατικών αλλαγών. Οι ίδιες χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που συνήθως κατά μέσο όρο έχουμε, παρατηρούν μια χρηματο, χρηματοπιστωτική ροή προς μεγαλύτερες πιο ε, ανθούσες ε, εκμεταλλεύσεις και τώρα έχουμε αντίθετα ε, στόχευση σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Με τις μεσαίες επιχειρήσεις το πρόβλημα είναι ότι είναι ο μέσο όρο ο δυσέβρετο, όπω σα είπα στην αρχή, γιατί δεν ανταποκρίνεται στην πλειοψηφία. Σε 5-10 χρόνια θα δούμε πώ θα αντιμετωπίσουμε αυτή την αίσθηση που έχουμε στι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει Οι αγροτικέ εκμεταλλεύσει. Επίση, περιβαλλοντικά μέτρα που δημιουργούν ε, επιπλέον απέτηση προσλήψεων και απασχόληση ή μέτρα ε, βελτίωση του βιωτικού επίπεδου, προκειμένου να παραμείνει και ο γεωργικός πληθυσμός στην Ήπεθρο, διαφοροποίηση των ε, δραστηριοτήτων, πρόθεση της ανανέωσης ε, της γεωργικής κοινωνίας, των αγροτικών κοινωνιών και επίσης κάποια σχέδια και προγράμματα για τους νέους γεωργούς που είναι πολύ σημαντικά για να προωθεί αυτή η ανανέωση των γενεών για να μπορέσουν οι νέοι μας γεωργοί να αναλάβουν τη σκητάλη από τους πιο ηλικιωμένος. Επίσης ζητήσαμε να ληφθούν υπόψη και ειδικά ζητήματα που αφορούν το φύλλο. Μέχρι στιγμής ε, τα θέματα του φύλλου δεν έχουν τύχει τη θέουσας προσοχής. Ακόμη το θέμα του φύλλου δεν φαίνεται ότι απασχολεί γενικότερα τον προβληματισμό για τη γεωργία στις χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης τουλάχιστον. Τώρα, ο ρόλος της Γεωργίας για το μέλλον στις εθνικές οικονομίες μειώνεται, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στην παραγωγικότητα αυξάνεται, στο λέω συνοπτικά, υπάρχει μεγάλος αριθμός μη μορφωμένων ηλικιωμένων γεωργών που εγκαταλείπουν το επάγγελμα. Βέβαια οι νέοι και ειδικευμένοι δεν ενθαρρύνονται να εισέλθουν λόγω των χαμηλών μισθών. Δύσκολο είναι να λάβει κανείς από τους γονείς την αγροτική μετάλλευση και επίσης δεν είναι αρκετά ελκυστικό το γεωρικό εισόδημα ή γεωρική δραστηριότητα. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε την προβολή της γεωργίας ώστε να γίνει πιο ελκυστική γεωρική δραστηριότητα για τους νέους. Υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση για γεωρική γη με μεγαλύτερη συγκέντρωση και μεγαλύτερη εντατικοποίηση Έχουμε ειδικέ τάσει, ιδιαίτερα στι ε, υπαίθριε καλλιέργειε που γίνονται πιο δημοφιλεί και στι ειδικευμένε ε, γεωργικέ εκμεταλλεύσει έχουμε μεγαλύτερου πόρου από το ανθρώπινο κεφάλαιο και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Αυτό είναι για μας ε, σημαντικό. Και τώρα, τι προτείνουμε για τις άμεσες ενισχύσεις θα πρέπει να βελτιώσουν την ικανότητα των γεωρικών εκμεταλλεύσεων να προσαρμόζονται καλύτερε στι οικονομικέ, περιβαλλοντικέ και κοινωνικέ αλλαγέ. Ωραία, ακούγεται αυτό, αλλά πώ θα γίνει. Θεωρούμε ότι περαιτέρω ενίσχυση τη περιβαλλοντική και κοινωνική πτυχή τη γεωργία ήταν κάτι θετικό. Επίση, η διευκόλυνση εντατικών συστημάτων παραγωγή με την ανακατανομή ή τον καθορισμό ανώτατου ορίου στην συνολική υποστήριξη. Τώρα, στο ό,τι αφορά την ανάπτυξη του πέθρου, θα πρέπει να βελτιώσει την ικανότητα των γεωργών να προσαρμόζονται καλύτερε οικονομικέ, περιβαλλοντικέ και κοινωνικέ αλλαγέ, με πιο ανταγωνιστικέ ε, γεωργικέ διαρθρώσει, με εξυγχρονισμό τη παραγωγή. Σημαντικό το θέμα του εξυγχρονισμού. Επίση, θα πρέπει να ενισχύσουμε την καινοτομία, τη μεταφορά τη τεχνογνωσία και τη συνεργασία. Ε, εξυγχρονισμό λοιπόν και καινοτομία, ε, θα πρέπει να διευκολύνουμε την, διαφοροποίηση με νέε προσοδοφόρες δραστηριότητε που δεν σχετίζονται με τη γεωργική εκμετάλλευση και τη διευκόλυνση της δημογραφικής ανανέωσης. Όλα αυτά περιστρέφονται κυρίως γύρω από την καινοτομία, γιατί όταν κάποιο είναι, κάτι είναι καινοτόμο, κάτι είναι υψηλή τεχνολογίας, όταν κάτι είναι σύγχρονο, τότε θα προσελκύσει τους νέους γεωργούς, τους νέους γενικά. Η καινοτομία λοιπόν είναι λέξη κλειδί για να προσελκύσουμε τους νέους γεωργούς. Και οι ευρωπαϊκή Εταιρικέ σχέση καινοτομία θα είναι ένα σημαντικό εργαλείο στο μέλλον. θα πρέπει να βάλουμε και τους γεωργούς στο παιχνίδι της καινοτομία. Έτσι θα βελτιωθεί η κατάσταση γενικά. Και αυτό το λέω όχι ως επιστήμονας, αλλά ως άνθρωπος που ενδιαφέρεται για τους γεωργούς και κυρίως τους νέους γεωργούς. Πιστεύω ότι η καινοτομία θα είναι το κλειδί για μια καλύτερη κοινή γεωργική πολιτική. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Ιωχάς. Περνάμε στον επόμενο καλεσμένο μας και να καλωσορίσω τους καλεσμένους της κυρίας Μαγκίνες τους ε, εκπροσώπους των Ιρλανδών Γεωργών. Ευχαριστούμε τους επισκέπτες της κυρίας Μαγκίνες που ήρθαν και τους καλωσορίζουμε θερμά. Παρακολουθείτε μαζί μας τις παρουσιάσεις των εμπειρογνωμών που καλέσαμε για να μας φωτίσουν με τις γνώσεις τους και να εμπλουτίσουμε τη συζήτηση. Εμφανίστηκε ο κύριος Λάιον στην αίθουσα. Τον καλωσορίζουμε. Θυμόμαστε ακόμη την θαυμάσια έκθεσή σας, κύριε Λάιον. Ευχαριστούμε λοιπόν και περνάμε στον επόμενο καλεσμένο, τον κύριο Σορεντίνο, τον καθηγητή Σορεντίνο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω Ιταλικά γιατί έλαβα κάποιες τέτοιες ε, οδηγίες λοιπόν. Έχω ετοιμάσει την παρουσίασή μου στα Ιταλικά. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Γεωργίας ε, και ε, τον Δ. Μάρτιν που μας σκέφτηκε για αυτή την παρουσίαση. Τώρα, μία εισαγωγή. Εμείς κάναμε μία ανάλυση οικονομικής φύσης κυρίως και επομένως οι συστάσεις πολιτικής ε, είναι συστάσεις που βασίζονται σε γενικές αρχές και όχι σε νομικές αρχές για την κατάρτιση διατάξεων δηλαδή. Όταν ε, ανέλαβα αυτό το έργο, αυτό το ερωτηματικό που έχουμε στο τέλος ε, του τίτλου μου προκάλεσε κάποια ανησυχία, κάποια ανησυχία για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα εδώ και πέντε χρόνια θέτει το πρόβλημα. Εδώ μάλλον και 50 χρόνια και παραπάνω θέτει το πώς θα απαντήσει σε αυτό το ερωτηματικό. Ήθελε να απαντήσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο στο παρελθόν για πολλά χρόνια, ενώ τα τελευταία χρόνια, όπως θα δούμε, έχουν αλλάξει οι τρόποι με τους οποίους ε, θέλει να απαντήσει σε αυτό το ερωτηματικό. Εδώ βλέπετε τη δομή της παρουσίασής μου. Εγώ θα αναφερθώ κυρίως στα σημεία 1, 3 και 5, καθώς τα σημεία 2 και 4 φαντάζομαι ότι είναι ήδη αρκετά γνωστά στην Επιτροπή σας. Περνάμε στο σημείο 1, το πεδίο εφαρμογή αυτής της ανάλυσης ξεκινά από μια προϋπόθεση ότι η κοινή γεωργική πολιτική μετακινείται προς ένα εντελώς καινούριο παράδειγμα, εντελώς καινούριος προς τη φύση του. Γιατί περνάμε από μια πολιτική δαπανών σε μια πολιτική ρυθμιστική στη διαδικασία μέσω της οποίας αυτή η πολιτική αναπτύσσεται. Δηλαδή από μία κεντρική παρέμβαση από πάνω προς τα κάτω, περνάμε τώρα στην προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Μία προσέγγιση η οποία ήδη χρησιμοποιείται ευρέως στις πολιτικές της αγροτικής ανάπτυξης και κυρίως αλλάζουν οι πρωταγωνιστές της πολιτικής ε, της ε, οργάνωσης των γεωργικών αγορών. Περνάμε από δημόσιους φορείς που σε κεντρικό επίπεδο δικούσαν και διαχειρίζονταν την κοινή οργάνωση αγοράς που ενώ τώρα περνάμε σε μια οργάνωση αγοράς που διοικείται κυρίω από τις οργανώσεις παραγωγών ή τι διαπαγγελματικέ οργανώσει. από ιδιώτες δηλαδή. Αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις. Όπως λέγαμε, ένα κεντρικό ρόλο διαδραματίζουν τώρα οι ιδιωτικές οργανώσεις. Δεν ε, βρισκόμαστε πλέον λοιπόν στη δημόσια σφαίρα, αλλά στη ιδιωτική σφαίρα. Έχουμε τις οργανώσεις των παραγωγών, τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και τις διεπαγγελματικές οργανώσεις. Στην ανάλυση αυτή εμείς ουσιαστικά θα αναλύσουμε το εργαλείο, το μέσο των οργανώσεων παραγωγών, γιατί θεωρούμε ότι προκειμένου να μπορούν να αναπτυχθούν διεπαγγελματικές οργανώσεις θα πρέπει να υπάρχουν παγιωμένοι συνομιλητές και οι οργανώσεις παραγωγών μπορούν να είναι για τους υπολείπους συμμετέχοντες στον τομέα συνομιλητές που μπορούν να τουτοποιηθούν πιο εύκολα και σίγουρα έχουν και καλύτερη αντιπροσώπευση. Αυτό το νέο παράδειγμα της παρέμβασης ε, στην οργάνωση των γεωργικών αγορών απαιτεί σίγουρα μία μεγάλη διαρθρωτική προσαρμογή η οποία σε αντίθεση με αυτό που βλέπουμε στο γεωργικό τομέα θα πρέπει να είναι ένα πολύ γρήγορο μέσο γιατί οι επιχειρήσεις ανάντι και κατάντι έχουν δυναμικές πολύ πιο γρήγορες από τις δυναμικές που χαρακτήριζαν τον αγροτικό τομέα. Μία άλλη πτυχή είναι η εξή. Δηλαδή, αυτό ο κεντρικό ρόλο των ιδιωτών στην οργάνωση των γεωργικών αγορών προκαλεί ανησυχίε για τον ανταγωνισμό στις γεωργικές αγορές και όλα αυτά φυσικά οδηγούν στο να χρειαζόμαστε μια συνεργασία μεταξύ ε, των αρχών που διέπουν την πολιτική ανταγωνισμού και των αρχών που διέπουν την γεωργική πολιτική. Διαχειρίζονται τη γεωργική πολιτική. Αυτή είναι μια πολύ σύντομη σύνοψη του τι αλλάζει στον γεωπιστιστικό κλάδο. Βλέπουμε ότι οι επιπτώσεις ε, στην οικονομία έχουν να κάνουν κυρίως ε, ε, με τον αριθμό των επιχειρήσεων και φυσικά δεν είναι κάτι που μπορούμε να παραβλέψουμε και φυσικά εξελίσσεται συνεχώς ο κλάδος και στρατηγικό ρόλο αναλαμβάνουν νέοι φορείς, νέοι πρωταγωνιστές οι οποίοι είναι εξαιρετικά εξωτερική ως προς τον κόσμο της αγροτιάς, όπως τα μίντια παραδείγματος χάρη. Αυτή η οικοδόμηση του κλάδου που αλλάζει τόσο βαθιά λόγω της ε, εισόδου αυτών των νέων παραγόντων είναι ένα γεγονός το οποίο μας οδηγεί σε μια απαραίτητη διαρθρωτική προσαρμογή και αυτό πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα. Εμείς στο σημείο αυτό έχουμε αναπτύξει ένα μοντέλο για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ποια μπορεί να είναι τα μέσα και ποια η αποτελεσματικότητα ορισμένων μέσων το να επαναξισορροπήσουμε την διαπραγματευτική δύναμη του κλάδου του γεωπιστητιστικού. Εμείς καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ορισμένους ορισμούς. Δηλαδή τι εννοούμε με την διαπραγματευτική δύναμη και με τη δύναμη της αγοράς. Η δύναμη της αγοράς σχετίζεται με μία δράση που έχει αποτελέσματα στο, επιπτώσει στο εμπόριο, στη ζήτηση και στην προσφορά όπως ε, είχαμε επίσης συνέπειες και στη συνολική ευημερία της οικονομίας. Όμως, αντίθετα, η διαπραγματευτική δύναμη ασκείται μέσω μιας απειλής. Της απειλής να αρνηθεί κάποιος τη συναλλαγή. Την απειλή να μην γίνουν σεβαστές κάποιες προϋποθέσεις, κάποιοι όροι. Αλλά όχι απαραίτητα τροποποιεί την ε, ισορροπία στην αγορά και στη ζήτηση. Παραδείγματο χάρη, εγώ μπορεί να περιορίσω την προσφορά για να προσπαθήσω να έχω πιο υψηλέ τιμέ. Έτσι λοιπόν, κάνω μία άμεση δράση. Ενώ στο μονοψώνιο εγώ περιορίζω τη ζήτηση ε, μίας ε, για να μπορώ να πληρώσω χαμηλότερη τιμή. Όμως την διαπραγματευτική δύναμη Εκεί δεν παίζω επί της τιμής και της ε, ποσότητας στην αγορά και στη ζήτηση, αλλά παίζω επί της απειλής του να μην πραγματοποιήσω τη συναλλαγή. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ενώ η εξουσία, τη δύναμη της αγοράς πάντοτε οδηγεί σε μία ε, απώλεια της ευημερίας η διαπραγματευτική δύναμη δεν οδηγεί απαραίτητα σε στρέβλωση του ανταγωνισμού, ούτε επιφέρει απαραίτητα μείωση της οικονομικής ευημερίας. Στο σημείο αυτό βλέπουμε ότι έχουμε σημαντικές συνέπειες γιατί όταν εμείς μιλάμε για διαπραγματευτική δύναμη οι ανησυχίε σε σχέση με τον ανταγωνισμό πρέπει να είναι πολύ διαφορετικέ σε σχέση με τι ανησυχίε που πρέπει να έχουμε στην περίπτωση που, που μιλάμε για δύναμη τη αγορά. Αν δούμε Βλέπουμε εδώ ότι η δύναμη της αγοράς ε, οδηγεί σε έλλειψη του προϊόντος, σε μη συνεργατική συμπεριφορά και επικεντρώνεται στο παιχνίδι τιμή ποσότητα. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά όμως που δεν χαρακτηρίζουν το γεπιστιστικό τομέα, ο οποίος αντιθέτως χαρακτηρίζεται από μια πολύ μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε μεγάλες ποσότητες, τεράστιες ποσότητες, από συντονισμό μεταξύ των ε, ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στα διάφορα στάδια του κλάδου και αποδράσεις που δεν έχουν να κάνουν μόνο με την τιμή και την ποσότητα, αλλά από μια πολυτομεακή ποικιλομορφία ε, των διαπραγματευτικών όρων. Όλα αυτά σημαίνουν ότι ο γεωπιστικός τομέας θα πρέπει να είναι ένα μοντέλο που θέλει να ενισχύσει τη διαπραγματευτική δύναμη και έτσι λοιπόν εδώ θα πρέπει να έχουμε ένα μοντέλο που να διαφυλάσσει και να αφορά την στη δύναμη και όχι τη δύναμη της αγοράς. Έτσι λοιπόν η πραγματική δύναμη είναι στο επίκεντρο της ανάλυσής μας γιατί εμείς θεωρούμε ότι όλα τα χαρακτηριστικά του γεωπιτοστικού κλάδου είναι χαρακτηριστικά τα οποία με πολύ καλό τρόπο ε, παρουσιάζουν την προστιθέμενη αξία του κλάδου μέσω της άσκησης της διαπραγματευτικής δύναμης. Αυτή είναι λοιπόν μια ταχεία απλούστευση του μοντέλου. Εμείς έχουμε τώρα εδώ ένα γεωργό και έναν αγοραστή. Βλέπετε εδώ την προστιθέμενη αξία αξία της ανταλλαγής και το εισόδημα που προκύπτει από αυτή την ανταλλαγή. Αυτό το εισόδημα μπορούμε να το αποσυνθέσουμε σε τρεις συνιστώσεις. Η μία συνιστώσα είναι ε, ουσιαστικά ε, αυτό που ο προμηθευτής ε, είναι το τμήμα της προσθέμενης αξία που ε, θα είχε το ίδιο ε, ο προμηθευτής. Δηλαδή είναι ένα εγκυμένο εισόδημα για τον Γεωργό, ακόμη και αν δεν γινόταν η συναλλαγή. Το κέρδος που θα είχε ο Γιώργος από, μια από ένα εναλλακτικό εμπόριο, το χάρη, με κάποιους άλλους τρόπους και με άλλους αγοραστές. Ενώ εδώ στην κόκκινη λωρίδα βλέπετε το disagreement payoff του αγοραστή. Δηλαδή το κέρδος που θα είχε ο αγοραστής αν ε, ουσιαστικά προμηθευόταν από άλλους γεωργούς και το ενδιάμεσο τμήμα είναι το περιθώριο της διαπραγμάτευσης. Με άλλα λόγια, τα δύο αυτά τα disagreement payoff καθορίζουν τις δύο διαπραγματευτικές θέσεις του γεωργού δηλαδή τη θέση της διαπραγμάτευσης του γεωργού και τη θέση διαπραγμάτευσης του αγοραστή. Σε αυτή την διάμεση πορτοκαλί λωρίδα βλέπετε το περιθώριο της διαπραγμάτευσης. Ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα από αυτή τη διαπραγμάτευση θα εξαρτηθεί από το εξής. Από τη διαπραγματευτική δύναμη. Δηλαδή, από τη δύναμη του ενός από τα δύο μέρη να καθορίσει τους κανόνες του παιχνιδιού, να καθορίσει τις ρήτρε όλης αυτής της ανταλλαγής, τους όρους της ανταλλαγής. Στο παράδειγμα μας, ε, τι να υποθέτουμε εδώ, γενικά υποθέτουμε ότι ένας αγοραστής ε, έχει ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη, δηλαδή έχει την ικανότητα να θέσει τους κανόνες του παιχνιδιού έναντι του Γιωργού. Έχει λοιπόν ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη, αλλά έχει και ισχυρή διαπραγματευτική θέση. Γιατί, Γιατί καθώς έχει απέναντί του πολλούς γεωργούς, έχει τεράστιες εναλλακτικέ δυνατότητες σε σχέση με τον Γεωργό, ο οποίος ε, ουσιαστικά δεν έχει μπροστά του πάρα πολλούς αγοραστές. Αν αυτή είναι η κατάσταση, ορίστε πώς ε, επιμερίζεται αυτό το κέρδος, το ποσοστό που πάει στον αγοραστή, το κόκκινο δηλαδή, και αυτό που πάει στο γεωργό, δηλαδή το κίτρινο μέρος. Επομένως, ε, ποιες ε, είναι οι διάφορες στρατηγικές. Είναι ουσιαστικά δύο. Είναι η διαπραγματευτική θέση των δύο μερών που εξαρτάται από τις εναλλακτικές που έχει το κάθε μέρος. Εγώ θα έχω μια καλύτερη διαπραγματευτική θέση στο βαθμό που θα έχω περισσότερες εναλλακτικέ σε σχέση με αυτή τη συναλλαγή. Αυτή είναι λοιπόν η διαπραγματευτική θέση. Όμως, όλο ε, σημαντικό στοιχείο που καθορίζει τη διαπραγματευτική δύναμη είναι η ικανότητα να ορίσει κάποιους του κανόνες του παιχνιδιού, τις διαπραγματευτικές ρήτρε, τους τρόπους μέσω των οποίων θα πρέπει να γίνει αυτή η συναλλαγή. Τώρα, στην επόμενη διαφάνεια, θέλουμε να δούμε το εξής ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος των οργανώσεων παραγωγών στο να εξισορροπηθεί η διαπραγματευτική δύναμη μεταξύ των δύο μερών. Εδώ, στο αποτέλεσμα, αυτό το αποτέλεσμα προέκυψε από μια κατάσταση όπου δεν έχουμε οργάνωση παραγωγού και έχουμε διάφορους γεωργούς και υποθέτουμε ότι υπάρχουν και λίγοι αγοραστές. Να δούμε τι συμβαίνει. Τη στιγμή που εμείς προσθέτουμε και οργανώσουμε τους ε, γεωργούς σε μια οργάνωση παραγωγού. Τι συμβαίνει. Έχουμε αποτελέσματα, επιπτώσεις και στη διαπραγματευτική δύναμη, αλλά στη διαπραγματευτική θέση. Γιατί αλλάζει η διαπραγματευτική θέση, γιατί η διαφωνία ε, το disagreement payoff των γεωργών μπορεί να αυξηθεί γιατί μια οργάνωση των παραγωγών υπό ορισμένε προϋποθέσεις έχει μεγαλύτερες δυνατότητες να βρει εναλλακτικές οδούς αγοράς από ό,τι θα μπορούσε να έχει ένας γεωργός μόνος του. Και σε επίπεδο οικονομίας κλίμακας. Δηλαδή, με άλλα λόγια τι λέμε. Λέμε ότι χάρη στην οργάνωση παραγωγών, οι γεωργοί μπορούν να έχουν περισσότερες εναλλακτικέ ε, αγοράς, μπορούν να θέσουν σε πορεία το προϊόν ε, σε διάφορες τυπολογίες αγοραστών και φυσικά αυτό αυξάνει τη διαπραγματευτική τους δύναμη. Βλέπετε όμως ότι επάνω το κόκκινο, η κόκκινη λωρίδα μειώνεται, γιατί μειώνεται η διαπραγματευτική θέση του αγοραστή. Γιατί ο αγοραστής ο οποίος πριν είχε πολλές εναλλακτικέ, γιατί είχε απέναντί του τόσους πολλούς παραγωγούς, τώρα θα έχει απέναντί του λίγες οργανώσεις παραγωγών και επομένως περιορίζονται οι εναλλακτικέ που έχει στη δυνατότητα που έχει στη διάθεσή του ο αγοραστής. Έχουμε λοιπόν αποτέλεσμα μια επίπτωση στη διαπραγματευτική θέση. Και βλέπετε ότι μετακινείται υπέρ των γεωργών. Υπάρχει και κάτι ακόμη. Θα δείτε ότι και η οριζόντια λωρίδα, το γαλάζιο δηλαδή, έχει μετακινηθεί προς τα πάνω στο περιθώριο διαπραγμάτευσης. Γιατί? έχει μετακινηθεί προς τα πάνω. Επειδή μια οργάνωση παραγωγών έχει τις προϋποθέσεις οικονομίας κλίμακας ε, και πεδίου που μπορούν να τις επιτρέψουν να υλοποιήσει μία σειρά υπηρεσιών αγοράς ακόμη καλύτερα από ένα μεμονωμένο παραγωγό που μπορούν να ενισχύσουν τη θέση των γεωργών ως προς το να θέσουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Δηλαδή να προσδιορίσουν ως αυτό που είπαμε διαπραγματευτική δύναμη. Αυτέ είναι λοιπόν οι επιπτώσεις. Έχουμε επιπτώσεις στη διαπραγματευτική θέση των γεωργών γιατί αυξάνονται ή πιθανές διέξοδοι στην αγορά. Υπάρχει ουσιαστικά και ένα αποτέλεσμα που περιορίζει τη διαπραγματευτική δύναμη του αγοραστή, γιατί δεν έχει ενωπιόν του τόσους πολλούς προμηθευτές, αλλά λιγότερους. Και Επίσης έχει επίπτωση και στη διαπραγματευτική δύναμη στο βαθμό που μία οργάνωση παραγωγών έχει περισσότερες δυνατότητες να επενδύσει στην αγορά και να αποκτήσει υπηρεσίες αγοράς για να μπορεί να συμμετάσχει ενεργά στον καθορισμό των κανόνων του παιχνιδιού. Προφανώς αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις. Μία επίπτωση έχει να κάνει με την ελάχιστη και αποτελεσματική διάσταση της οργάνωσης παραγωγών. Και πολλές μικρές οργανώσεις παραγωγών ε, τελικά δεν μπορούν να καταλήξουν σε αυτά τα αποτελέσματα που είδαμε παραπάνω. Γιατί συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει γιατί πολλές μικρές οργανώσεις αγοράς δίνουν πολλές εναλλακτικέ ευκαιρίες στον αγοραστή και επομένως δεν περιορίζεται η κόκκινη λωρίδα τόσο πολύ. Γιατί οι μικρές οργανώσεις παραγωγών δεν ε, αποκτούν εύκολα αυτή την οικονομία κλίμακας για να παράσχουν μια σειρά υπηρεσιών αγοράς που να τους επιτρέψουν να βελτιώσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη. Και φυσικά αυτή η ελάχιστη διάσταση έχει στρατηγική πολιτική σχετικότητα και φυσικά θα πρέπει να αξιολογηθεί πολύ προσεκτικά σε σχέση με τη δομή της αγοράς ανάντι. Εμείς κάναμε αυτό το μοντέλο και κάναμε και μια σειρά προσωμιώσεων. Παραδείγματος χάρη σε μια κατάσταση όπου έχουμε ένα μόνο αγοραστή, αν οι γεωργοί θέλουν να αυξήσουν το ποσοστό του της αξία στην αναλλαγή κατά 20% θα πρέπει τότε να ομοδοποιηθούν όχι πάνω από έξι οργανώσεις παραγών. Δηλαδή πρέπει να έχουμε όχι περισσότερο από 6 οργανώσεις παραγωγών έναντι ενός αγοραστή για να έχουμε 20% αύξηση προσθεμένης αξίας του Γιωργού. Αν αντίθετα έχουμε τρεις αγοραστές, τότε θα αρκούν 10 οργανώσεις παραγωγών για να φτάσουμε στην αύξηση του 20% της προσθέμενης αξίας που αντιστοιχεί στο Γιωργό. Εμείς στο έγγραφο έχουμε και μια σειρά προσωμιώσεων, έχουμε και γραφήματα και θα δείτε ότι η κατάσταση της αγοράς ανάντι επηρεάζει πάρα πολύ την ε, επιλογή σε σχέση με την ε, ελάχιστη διάσταση που πρέπει να έχουμε στις οργανώσεις παραγωγών έτσι ώστε να μπορούν να αυξήσουν η παραγωγή την προστιθέμενη αξία που αντιστοιχεί στους γεωργούς. Και εδώ λοιπόν ε, έχουμε την ελάχιστη διάσταση που είναι ένα θέμα ε, κλειδί. Ένα άλλο θέμα έχει να κάνει με τις επενδύσεις των οργανώσεων παραγωγών στο να δημιουργήσουν εναλλακτικές οδούς αγοράς. Όσο περισσότερο μπορεί η οργάνωση παραγωγών να δημιουργήσει τέτοιε εναλλακτικέ οδού αγορά, τόσο περισσότερο θα αυξηθεί η διαπραγματευτική τη θέση και επομένως το ποσοστό της προσθέμενης αξίας της συναλλαγής. Μια άλλη στρατηγική μεταβλητή είναι η ικανότητα της οργανώσεως ε, παραγωγών να αποκτήσει νόμιμες και εμπορικές υπηρεσίες για να αντιμετωπίσει κάποιες αθέμητες εμπορικές πρακτικές. ακόμη και αν έχουν σημαντικό ρόλο, παραδείγματο ε, χάρη στην ε, πρωτοβουλία της ε, λυσίδας εφοδιασμού. Σήμερα, βέβαια, οι γεωργοί εκπροσωπούνται πολύ λίγο εκεί. Ίσως να μπω κατευθείαν στα συμπεράσματα. Τα έχετε εδώ. Λοιπόν, εμείς έχουμε κάποια συμπεράσματα για την αποδοτικότητα των οργανώσεων παραγωγών, για την αποτελεσματικότητα, για το σχεδιασμό αυτών των οργανώσεων, για τα κέρδη της αποδοτικότητας και για τη στρατηγική των οργανώσεων παραγωγών. Καταρχήν, τι μπορούμε να πούμε μπορούμε να πούμε ότι η συγκέντρωση της προσφοράς ε, που γίνεται από τις οργανώσεις παραγωγών δεν επιφέρει απαραίτητα στρέβλωση του ανταγωνισμού και ούτε βλάπτει τη λειτουργία της αγοράς. Όμως αυτό εξαρτάται πάρα πολύ από την διαχείριση, τη διακυβέρνηση των οργανώσεων παραγωγών. Υπάρχουν μία σειρά ε, όρων που πρέπει να σεβαστούν οι οργανώσεις παραγών προκειμένου να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη αλλά να μην, να μην μεταμορφώσουν τη διαπραγματευτική δύναμη σε δύναμη της αγοράς. Και ποιες είναι αυτές οι ενδείξεις. Κυρίως οι οργανώσεις παραγωγών θα πρέπει να έχουν ελευθερία εισόδου-εξόδου, θα πρέπει η οργάνωση παραγωγών να δεκτεί κάθε ποσότητα που θέλουν να συνεισφέρουν τα μέλη της στην οργάνωση, που θέλουν δηλαδή να διαπραγματευτούν μέσω της οργάνωσης παραγωγών. Ουσιαστικά αυτές είναι οι δύο προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητα. Εδώ είπαμε ότι αυτό εξαρτάται από πολλά πράγματα. Σίγουρα εξαρτάται από τη δομή της αγοράς, ανάντι και κατάντι. Δηλαδή πόσο συγκεντρωμένη ε, είναι η παραγωγή ανάντι και κατάντι. Γενικά η συγκέντρωση της προσφοράς από την πλευρά της οργάνωσης παραγωγών έχει θετική επίπτωση στη διαπραγματευτική δύναμη των γεωργών και αρνητική επίπτωση στη διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών. Όμως η διάσταση αυτών των αποτελεσμάτων συνδέεται στενά με την συγκέντρωση ανάντι και κατά Αν ανάντι είναι ε, υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση στον τομέα, οι οργανώσει παραγών θα πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλε για να μπορούν να είναι αποτελεσματικέ σε κάποιο βαθμό. Έχουμε συμπεράσματα για το σχεδιασμό, για τη μορφή που πρέπει να έχει μια οργάνωση παραγωγών. Μια πολύ μικρή οργάνωση πιθανότατα θα είναι αποτελεσματική στο να βελτιώσει τη διαπραγματική δύναμη των γεωργών. Προφανώς, όπως έλεγα, στην ε, βεθμονόμηση της διάστασης οργάνωση παραγωγών και, στην, στο μερίδιο της αγοράς είναι πολύ σημαντικό το επίπεδο συγκέντρωσης ανάντι και κατάντι. Είπα, αν υπάρχει πολύ μεγάλη συγκέντρωση, των επιχειρήσεων, ανάντι και κατάντι, το μερίδιο της αγοράς, ε, της οργάνωσης παραγωγών θα πρέπει να είναι αρκετά υψηλό. Θα πρέπει. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλο μερίδιο. Μία άλλη πτυχή, στην οποία δεν αναφέρθηκα πολύ, αλλά αναφέρεται εκτενώς των έγγραφο, είναι το θέμα της αποδοτικότητας στη σημερινή νομοθεσία αποτελεί προϋπόθεση για την παρέκκληση για τις παρεκκλήσεις ως προς τον ανταγωνισμό. Όμως εδώ θα έλεγα ότι πρέπει να το δούμε περισσότερο ως ευκαιρία, όχι ως προϋπόθεση. Γιατί στο βαθμό που οι οργανώσεις παραγωγών αυξάνουν την αποτελεσματικότητά τους, την αποτελεσματικότητά τους, μπορούν να έχουν μία συμφωνία win-win όπου θα υποφεληθούν και οι οργανώσεις παραγωγών και οι διακαταναλωτές αλλά και οι αγοραστές. Όμως για να υπάρχουν θετικά αποτελέσματα για τις οργανώσεις παραγωγών, οι οργανώσεις αυτές θα πρέπει να έχουν μια διαπραγματευτική δύναμη μεγάλη. Και η τελευταία πτυχή έχει να κάνει με τις στρατηγικές αγοράς των οργανώσεων παραγωγών. Είπαμε ότι μια πολύ σημαντική πτυχή είναι αυτή της διαπραγματευτικής θέσης. Η διαπραγματευτική θέση των παραγωγών και σε ποιο βαθμό έχουν πολλές εναλλακτικές να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Επομένως, τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αφήσουμε στις οργανώσεις παραγωγών τη μέγιστη βιλξία ως προς το να βρουν τις καλύτερες διόδους, τους καλύτερους διάβλους στην αγορά. Ίσως εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε και μία υπόθεση, μία πρόταση. Δηλαδή να μην περιοριστούν οι οργανώσεις παραγωγών σε ένα και μόνο προϊόν. Τέλειωσα, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά. Πανεπιστημιακή διάλεξη. Ο κύριος Χανιώτης τώρα. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Uh, thank you, Chairman, and thanks also for... Uh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους καλεσμένους για τις ε, παρουσιάσεις. Θα είμαι λακωνικός, θα σας απασχόλησω πολύ. Θα σας εξηγήσω πού επικεντρωνόμαστε εμείς σε θέματα διαρθρωτικών προσαρμογών. Γιατί οι διαρθρωτικές προσαρμογές έχουν ε, σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση της ΚΑΠ. Είναι γεγονός βέβαια στη Γεωργία παντού στον κόσμο, άσχετα από τις πολιτικές που εφαρμόζονται, την έλλειψη πολιτικών. Είναι περίπλοκο και ασύμετρο φαινόμενο και ως προς τις ε, μεθόδους παραγωγούς, ως προς τα κράτη-μέλη, αλλά και ως προς τις καταστάσεις στις διάφορες περιφέρειες που έχουμε διαφορετικούς τρόπους παραγωγής μεταξύ των παραγωγών. Και σε μεγάλο βαθμό έχουμε κάποιες μακροεξελίξεις ε, εκτός της γεωργίας που επηρεάζουν τις διαφορετικές αυτές αλλαγές και επηρεάζονται επίσης από μικρο συμπεριφορές. Και αν δούμε τις λεπτομέρειες ε, των δεδομένων για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, διαπιστώνουμε ότι για την ίδια παραγωγή, για τα ίδια χαρακτηριστικά, με πολύ διαφορετικό τρόπο ανταποκρίνονται οι μεμονωμένοι γεωργοί. Στα νεότερα κράτη-μέλη είχαμε όντως ταχύτερο ρυθμό ε, διαρθρωτικών προσαρμογών στη γεωργία. Α, κάτι αναμενόμενο, γιατί είχαν πολύ μικρότερη περίοδο προσαρμογής και είχαν και ταχύτερους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης γενικώ. Αυτό όμως που είναι πιο ενδιαφέρον είναι ότι εντός και των 15 χωρών, των 10 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε διαφορές, μεγάλες διαφορές στις διαφορετικές αλλαγές. Ο δημογραφικός παράγων παίζει σημαντικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Η γύρανση του γεωργικού πληθυσμού. Και εκεί υπάρχουν διαφορές όμως. Και ίσως ε, το μόνο κοινό στοιχείο είναι η μεροληψία ως προς το φύλλο. Επίσης, το καλοκαίρι οργανώσαμε ένα εργαστήριο, πέρυσι το καλοκαίρι μάλλον, στο περιθώριο της ΕΚΣΠΟ, της Διεθνούς Έκθεσης του Μιλάνου, για να δούμε ε, τις συνέπειες που έχει το μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και το αποτέλεσμα, το πόρισμα αυτής, αυτού του εργαστηρίου ήταν ε, δεν επηρεάζει το μέγεθος στην αποτελεσματικότητα της ε, συμπεριφοράς του γεωργού. Γιατί έχουμε αποδοτικέ ή μη απόδοτικέ γεωργικέ ε, εκμεταλλεύσεις, φιλοπεριβαλλοντικές ή όχι, άσχετα με το μέγεθός τους. Σε ό,τι αφορά τι συνέπειε της πολιτική, Κάνουμε μια επικαιροποίηση της ε, έκθεσης για το 2020 που πριν από 10 χρόνια ξεκίνησε το Πανεπιστήμιο του Βάγκενιγκεν για να το φέρουμε στα σημερινά επίπεδα τιμών. Η μελέτη έλεγε ότι η τοποθεσία ασκούσε μεγαλύτερο ρόλο από ότι το μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης. Ακόμη και ελλείψη πολιτικών, ακόμη και ελήψη κοινή γεωργικής πολιτικής, θα είχαμε ταχύτερες διαρθρωτικές προσαρμογές, με μεγαλύτερη συγκέντρωση στις πιο ανταγωνιστικές ε, περιφέρειες και μεγαλύτερη εγκατάλειψη γεωργικών γεών στις περιφερειακές ή πιο απόμακρες περιοχές. Και παρά την πρώτη ομιλία, εμείς δεν θεωρούμε ότι υπήρχε μία ε, θετική διάκριση υπέρ των μεγαλύτερων γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Στην αρχή το επίπεδο παραγωγής ε, ε, έπαιζε ρόλο. Όταν είχαμε αποσύνδεση με το πάγωμα των πληρωμών, τότε είχαμε μία πιο ουδέτερη κατάσταση. Βέβαια δεν υπάρχει ομοιομορφία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι πιο περίπλοκο το θέμα και σίγουρα δεν υπάρχει θετική διάκριση υπέρ των μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Ε, αναλαμβάνω και το μέγεθο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων δεν είναι το ίδιο στι διάφορε παραγωγέ. Άλλο να μιλάμε για εντατική γεωργία απορροκυπευτικών και το μέγεθο εκεί, και άλλο να μιλούμε για κτηνοτροφία. Και τα περισσότερα κράτη-μέλη επέλεξαν να υιοθετήσουν την ίδια πολιτική, την κοινή ιδιωτική πολιτική, με διαφορετικό τρόπο, με περιφερειακά μοντέλα, με ιστορικό μοντέλο, με συνδεδεμένε ή αποσυνδεδεμένε ενισχύσει. Τώρα, για να κάνουμε και κάποιε προβλέψει, να προλάβουμε το μέλλον, η επιδείνωση των διαπραγματευτικών όρων ε, στις, ε, στα γεωργικά προϊόντα όπου οι τιμές των γεωργικών προϊόντων αυξήθηκαν το 1 δέκατο των τιμών των λοιπασμάτων των ενεργειακών προϊόντων, προϋποθέτει ανάγκη να επικεντρωθούμε σε τρία πράγματα που θα εξαρτήσουν στο μέλλον τις διαρθρωτικές προσαρμογές. Καταρχήν, το quiz του κόστους που αντιμετωπίζουν, που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί και θα πρέπει να δούμε τις διαφορετικές ε, ε, προκλήσει σε άλλα τύπου προϊόντων. Και δεύτερον, οι προκλήσει από τι αλλαγέ τη κλιματική και του περιβάλλοντο απαιτούν την ανάπτυξη γεωργία βασισμένη στη γνώση και διαχείριση τη υγή. Αυτό σημαίνει διαφορετικέ προκλήσεις αναλόγως, αναλόγως της ηλικίας του παραγωγού, της τεχνολογίας που χρησιμοποιεί, την κατάρτιση, τις συμβουλές που θα έχει στη θέση του, τα σχετικά με τη μεταφορά τον της γνώσης και βέβαια την νοοτροπία. Και εν τέλει είναι πολύ σημαντικό, είναι άκρο σημαντικό δεδομένων των ε, αλλαγών πολιτικής ε, που μπορεί να βοηθήσουν στην κατεύθυνση της μίας της ελευθερωτικής αλλαγής. Πρέπει να υπάρχουν σαφείς ιδέες για τις συνέπειες των μέτρων πολιτικής που μπορεί να προκύψουν, δηλαδή είτε εστιαζόμενος κανείς στις τιμές, είτε εστιαζόμενος στο εισόδημα, γιατί δεν είναι ουδέτερος προς τις γενικές συνέπειες. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, πριν να περάσουμε στις ερωτήσεις των βουλευτών, θα ήθελα να καλωσορίσω εδώ και τους εκπροσώπους Ιταλών Γεωργών που έχει προσκαλέσει ο συνάδελφος Τεντσούλα. Σας καλωσορίζω λοιπόν όλους και χαίρομαι που είστε εδώ μαζί μας για να παρακολουθήσετε τη συζήτησή μας. Χαίρομαι που μπορείτε να ακούσετε και τις αυτές, θεματολογικές αυτές ε, τοποθετήσεις των ειδικών μας ε, έχουν να κάνουμε δύσκολα ζητήματα όπως αυτά των ερθωτικών αλλαγών. Σας καλωσορίζω λοιπόν και τώρα μπορούμε να ακούσουμε, όχι να αρχίσουμε μια συζήτηση θα έλεγα, αλλά να ακούσουμε τις τοποθετήσεις των βουλευτών. Παρακαλώ, ο κύριος Ντες Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ θερμά τους ομιλητές μας για τις παρουσιάσεις τους. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες και οι αξιολογήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω αν συμφωνείτε μαζί μου ότι δεν υπάρχει μία απόλυτη συνταγή για τη γεωργία στην Ευρώπη. Έχω δώσει στατιστικές της Ρουμανίας όπου 29,1% των, ε, του ενεργού πληθυσμού εργάζεται ε, στη γεωργία, 12,5% ε, στην Πολωνία, 1,2% στο Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα είναι σχετικά μικρός ορισμένος χώρος το ποσοστό του ενεργού πληθυσμού που ασχολείται με τη γεωργία και θα ήθελα εδώ να πω μια και έχω παρακολουθήσει την ε, εξέλιξη του γεωργικού τομέα από το 1961 είχαμε στην περιοχή μου 65 ε, γεωργούς και έναν τσαγκάρι και έναν ακόμη εργαζόμενο σε άλλο τομέα. Δηλαδή δεν υπήρχε άλλη γεωργική δραστηριότητα. Πέραν αυτού άρχισαν σιγά σιγά να κερδίζουν μέρος του εισοδηματό τους γεωργοί και σε άλλους τομείς. Και τώρα έχουμε και δύο γεωργούς που ασχολούνται και με την ε, πυρόσβεση. Έχουμε 20 γεωργούς οι οποίοι εργάζονται και συμπληρώνουν το εισόδημά τους πέραν της γεωργίας. Όμως σε σχέση με το 1981 έχουμε περισσότερο εργατικό δυναμικό που απασχολείται στις εκμεταλλεύσεις γιατί χρειάζεται για να διαφυλαχθεί η λειτουργία της εκμετάλλευσης, η εγκατάσταση μιας νέας εκμετάλλευσης ε, και επιπλέον προσωπικό. Είναι περισσότερες οι θέσεις εργασίας που έχουμε λοιπόν στη Γερμανία, στην Γεωργία, στη Γερμανία, στην περιοχή μου από ότι το 1981. Μεγάλες συστήσεις ή προβλήματα δεν υπήρξαν. Όλα επελήφθησαν όποτε υπήρξαν ε, με τις κοινωνικές, με τις λογικές διαπραγματεύσεις και θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχουν διαφορετικές εικόνες της γεωργίας ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή και γι' αυτό δεν μπορεί να υπάρξει μία μόνο συνταγή για την ε, επιτυχία της γεωργικής δραστηριότητας. Πρέπει πάντα να κοιτάμε τις εταιρείες συνθήκες και κάτι ακόμη θα ήθελα να επισημάνω σε σχέση με τον στόχο για την ανάπτυξη μιας πιο παραγωγικής γεωργικής οικονομίας. Νομίζω ότι μπορούμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα, όπως είπατε και εσείς, αλλά ταυτόχρονα θα ήθελα να πω ε, για έναν συνεταιρισμό και τον πρόεδρό του, συνεταιρισμό γαλακτοπαραγωγικό, που είχαμε ουσιαστικά το μονοπόλιο με δύο ε, συνεταιρισμού στη Γερμανία και δύο μόνο είδη τυριού που παρήγαγαν. Παρήγαν καλύτερα. Τώρα έχουμε από ένα γειτονικό κράτος ε, εξαγωγέα, ο οποίος έριξε στην αγορά 800 τόνους διαφορετικού τυριού και κατέστρεψε όλη αυτή την ισορροπία. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι δεν μπορούμε μόνο με την ε, ισχύουσα θέση, με, την, με μια ισχυρή θέση στην αγορά να πούμε ότι έχουμε λύσει τα προβλήματα, διότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να προκύψει μια νέα συνθήκη η οποία ανατρέπει τρέπει τις αυτέ. αυτές. Δεν θέλω να σας καθυστερήσω περισσότερο βεβαίω και άλλοι συναδελφοί είναι εδώ για να διατυπώσουν τι ερωτήσει του, Ωστόσο, πρέπει να συστήσουμε εντατικά πιστεύω Πώ σε χώρε όπου υπάρχουν πολλές, πολύ μικρές εκμεταλλεύσεις και είχα αναλάβει ο καθήκον να μελετήσω και στατιστικές ε, για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 70% των εκμεταλλεύσεων στην Ευρώπη είναι μικρότερες των 5 εκταρίων. Αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη λοιπόν όταν κοιτούμε στοιχεία του 80-81 του που μας αναφέρατε ότι άρχισαν να συλλέγονται με 30 ώρες εργασίας για την συγκομιδή γενικά εκμετάλλευση και συγκομιδή ενό εκταρίου και τώρα μπορούν να αρκούν 20 ώρε νομίζω ότι ασφαλώ θα υπάρξουν διαρθρωτικές αλλαγέ για τη εισαγωγή τη νέα σύγχρονη τεχνολογία, επιτρέπει την εκμετάλλευση ταχύτερα μεγαλύτερων ε, εκτάσεων. Και νομίζω ότι θα πρέπει ταχύτατα να δώσουμε απαντήσει και σε σχέση με την ε, συμπληρωματική οικονομική δραστηριότητα που μπορεί να επιτρέψει συμπληρωματικό εισόδημα για το Γιώργο. Ο Πρόεδρος. Άλλος ομιλητής παρακαλώ, κύριος Δεκάστρο. Sí. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τους εμπειρογνώμονες και οι τρεις παρουσιάσεις ήταν ενδιαφέρουσες και φυσικά πολύ πλούσιες και θα μας δώσουν πολύ τροφή για σκέψη. Σίγουρα το θέμα των διαφορετικών αλλαγών είναι πολύπλοκο και είναι διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν. Και μάλιστα ο κύριος Χανιώτης το υπενθύμησε ανάλογα με την τοποθεσία μπορεί να αλλάξει και η ταχύτητα των διαφορετικών αλλαγών. Όμως εγώ θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση που μου ήρθε στο νου ακούγοντας και τον κύριο Ντες ε, όταν αναφερθήκε στη χώρα του. Εμείς ε, επί της ουσίας έχουμε μία, ένα μέγεθος ε, επιχείρησης πολύ μικρό. Αν συγκρίνουμε την Ευρώπη με τις υπόλοιπες περιοχές του κόσμου, τη Βόρεια Αμερική, την Αυστραλία, το πρόβλημα είναι αυτή η βραδύτητα με την οποία γίνονται οι διευθυντικές αλλαγές, πώς μπορεί να βελτιωθεί μέσω ε, διάφορων ε, μέσων που προσφέρονται, όπως το χάρη, μέσω των οργανώσεων παραγωγών. Εμείς στην Ιταλία Παραδείγματο χάρη έχουμε πάρα πολύ μικρές γεωργικές επιχειρήσεις, όμως η οργανωτική τους ε, απόδοση είναι πάρα πολύ καλή και είναι ανταγωνιστικές στην αγορά. Και ο συνάδελφο Τόρφμαν το ξέρει πολύ καλά. Μιλάμε, παραδείγματο χάρη, ε, για 1,5 εκτάριο ε, κατά μέσο όρο είναι η έκταση της επιχείρησης, της εκμετάλλευσης και όμως ε, κατορθών να εξαγάγουν και προϊόντα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Έτσι λοιπόν, πόσο τα μέσα ε, τις διάρθρωσης προσφορές μπορούν να μας κάνουν να επιταχύνουμε λίγο αυτές τις διαρθρωτικές αλλαγές. Σας ευχαριστώ και πάλι συγχαρητήρια. Ο κύριος Ευχαριστώ. Έχω τρία σχόλια, τρεις κατηγορίες σχολείων για τους τρεις καλεσμένους. Από τον πρώτο εμπειρογνώμονα από τις κατοχώρες. Είπατε ότι η τάση είναι να μεγαλώνουν οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Υπάρχει όμως και άλλη δυναμική τάση. Ε, για φανταστείτε ένα γεωργό που έχει δύο ε, γιους που απασχολούνται στη γεωργική εκμετάλλευση και πάνε καλά. Όταν τα δικά τους παιδιά, τα εγγόνια δηλαδή, ε, θέλουν να αναμειχθούν. Εκεί δημιουργούνται προβλήματα. Και συνήθω η λύση είναι η διαίρεση τη γεωργικής εκμετάλλευση. Οπότε διαιρείται η μία μεγάλη γεωργική εκμετάλλευση σε τρει, τέσσερι, πέντε αγροτικέ Έχουμε τέτοια παραδείγματα και είναι μια αντίστροφη δυναμική δηλαδή, μια τάση αντίστροφη αυτή. Οι μικρε αγροτικε εκμεταλλεύσει ουσιαστικά στηρίζουν τι μεγαλε και μπορούν να το κάνουν. Για παράδειγμα, για, τις, ε, για τους σπόρους, η ε, μικρή ε, γεωργή είναι έτοιμος ε, να προσέξει για τον πολλαπλασιασμό του αναπαραγωγικού υλικού. Γιατί οι σπόροι είναι πολύ ακριβοί και η προσοχή στη λεπτομέρεια που έχουν οι μικροί γεωργοί είναι μεγαλύτερη από ότι οι μεγάλοι. Γιατί οι μεγάλοι γεωργοί απασχολούνται με τα βάσανα των μεγάλων εκμεταλλεύσεων που έχουν και ο μεγάλος γαλακτοπαραγωγός επικεντρώνεται κυρίως ε, στον, ε, στην παραγωγή γάλακτος. Ενώ η μικρή παραγωγή δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στον παραγωγικό υλικό και ίσως ε, μερικές φορές οι μεγάλες εταιρείε, οι μεγάλε γεωργικέ άλλα αναθέτουν μερικά τμήματα αναζήτησης και προσοχή τα μέρες μικρότερε. Επίση, μιλήσατε, η δεύτερη ομιλήτρια μας μίλησε και για τη δυσπιστία ίσως ήταν κατάλοιπο τον, το προηγούμενο καθεστώτος. Το 1970, όταν ήμουν απλός φοιτητή, έμαθα στο σχολείο ότι επίκειτο κίνδυνο. Ο μέσος όρος ε, ηλικίας ήταν 58 έτη για τους γεωργούς. Και αν η κυβέρνηση δεν αναλάβανε άμεσα μέτρα για να εμπλέξει και νεότερους, ε, θα το μεγάλος κίνδυνος με ηλικιωμένου γεωργού που θα εγκατέλειπαν τι γεωργικέ εκμεταλλεύσει. Και η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα. Και πριν από ένα χρόνο Κάποιο μου είπε ότι η μέση ηλικία των γεωργών είναι 57 για τους Άγγλους γεωργούς και αν δεν κάνουμε τίποτα άμεσα θα μας περιμένει μεγάλη καταστροφή. Μην ανησυχείτε λοιπόν. Ε, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Γενικώ ο κόσμο ξέρει πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να βγει στη σύνταξη. Επίση είπατε δεν είναι και πολύ σεξι γεωργία, δεν είναι πολύ ελκυστική. Δεν συμφωνεί η Συνομοσπονδία Νέων Γεωργών τη Μεγάλη Βρετανία με το σχόλιο ότι δεν είναι ελκυστική η γεωργία για του νέου. Τώρα για τον Ιταλό καλεσμένο μας. Πολλά είπατε που μπορεί να είναι σωστά στη θεωρία, αλλά στην πράξη δεν ευσταθούν. Για παράδειγμα, η διαπραγματευτική ισχύ. Όντω, έχουμε οργανώσει παραγωγών, αλλά θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλες για να έχουν τέτοια ισχυρή διαπραγματευτική ισχύ και να πείσουν τα μέλη του να αντισταθούν και να δεχτούν μόνο μεγάλε πολλέ τιμές. Γιατί μερικοί εκμεταλλεύονται από την αύξηση των τιμών, γιατί οι βασικοί ανταγωνιστές δεν κάνουν τίποτα. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες και να βρεθούν κερδισμένοι όχι κατάλληλοι άνθρωποι. Επίσης, πώς θα σταματήσουμε την παραγωγή. Δεν μπορεί να πει κανείς στην κότα να σταματήσει να γεννά ή στην Αγελάδα να σταματήσει να παράγει γάλα. Και είναι πολύ πιο δύσκολο να το εφαρμόσουμε στην πράξη. Θεωρία ακούγεται καλά, αλλά στην πράξη είναι δυσεφάρμοστο. Και αν πείτε, εντάξει, έχουμε μεγάλες, ε, τεράστιες οργανώσεις παραγωγών και αυτές μπορούν να απεργήσουν ή να κατεβάσουν το ρόλο, τότε θα είχε όντω μεγάλη διαφορά στη διαπραγματευτική σχήμα. Πάντω, στην Μεγάλη Βρετανία έχουμε τέτοιο, τέτοιο δίκαιο ανταγωνισμού που θα καταστούσε αδύνατο κάτι τέτοιο. Θα καταστούσε αδύνατο κάτι τέτοιο. Οπότε, αν είναι κανείς στη λάθος πλευρά του στρατοπέδου είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και στην Αργεντινή ε, κατέβηκαν σε απεργία οι Γεωργία, αλλά αφού είχαν ολοκληρώσει το θερισμό και αποθήκευσαν το καλαμπόκι για να καταφέρουν να ανεβάσουν τις τιμές. Αλλά αυτό ισχύει μόνο για τις αρρώσιμες καλλιέργειες όταν ήδη τις έχουν αποθηκεύσει, έχουν προβεί στο θερισμό και έχουν αποθηκεύσει τον καρπό. Ευχαριστώ. Κύριε Σουαζό. Oui, merci, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα το να υποστηρίξουμε το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Μοντέλο του 21ου αιώνα μέσω της ε, ΚΑΠ ε, είναι πραγματικά παράλογο. Απλώς ε, η ΚΑΠ καταστρέφει αυτή τη γεωργία και ξέρετε ότι εδώ και καιρό η κατάσταση στην Ευρώπη αλλά και στη Γαλλία υποβαθμίζεται κυρίως μέσω της απορρίθμισης της παραγωγής και επίσης και από το ρωσικό εμπάργκο και από τον αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών και το πρασίνισμα της ΚΑΠ με ε, κάποια πολύ περιοριστικά μοντέλα, το χάρη, εγώ που είμαι γεωργός όπως γνωρίζετε εδώ και χρόνια βιώνω αυτή την κατάσταση. Η εκμετάλλευσή μου ε, πραγματικά βιώνει τα αρνητικά αποτελέσματα της ε, ΚΑΠ ε, και αναφέρθηκε η απλούστευση της ΚΑΠ. Όμως θα μπορούσε ουσιαστικά αυτό που να κάνει είναι να απελευθερώσει τους αγρότες από τη γραφειοκρατία και από τα εμπόδια της δίκησης και μιλώ ακριβώς για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο δεύτερο πυλώνα. Επίσης ε, ε, τελικά νομίζω ότι τα κράτη αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιστούν πάρα πολύ ε, δύσκολη την εργασία των Γεωργών. Νομίζω ότι λείπει πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα από την δική σας κοινή γεωργική πολιτική. Σας ευχαριστώ. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik heb een, eh, een vraag aan... Eh, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση για τον κύριο Φαντομπλούχο από το Βάχνιγκεν. Κοιτάμε για τη γεωργία, μιλούμε για τις κατοχώρες, αν ξεπίθουν και άλλοι τομείς να συζητήσουμε. Ερωτώ λοιπόν τι γίνεται με τις, οικονομικ... με τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις σε σχέση με τις μηχανικής κλίμακας. Ποια είναι η κατεύθυνση. Ο Πρόεδρος. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τη γερμανική διερμηνία. Παρακαλώ, θα είχατε καλοσύνη να ξεκινήσετε από την αρχή. Ε, να τα πω στα γερμανικά λοιπόν. Να τα πω, όχι μάλλον, στα ολλανδικά τελικά. Είναι σαφές λοιπόν ότι μιλάτε για έξι, πέντε cents του ευρώ για το γάλα, μιλούμε για το χείριο. Είδατε την παρατήρηση του κυρίου Ντές για τη Γερμανία. Ρωτώ λοιπόν ποια είναι η θεωρή σας για το μέλλον τη γεωργίας στην Ευρώπη, αλλά και ειδικότερα τη κατοχώρες σχέση με τι οικογενικές εκμεταλλεύσει. Και θα ήθελα και κάποιες απόψει. γιατί πολλέ θα είναι οι οικογενειακέ εκμεταλλεύσει κατοχώρες οι οποίε μπορούν να επηρεαστούν. Ο κύριος Δόρφμαν, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για τον καθηγητή Σορεντίνο. Θέλω να, να, θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Σορεντίνο. Πιστεύω ότι είναι σαφές ότι η οργάνωση παραγωγών επιφέρει μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη. Αυτό δεν ε, οφείλεται μόνο στις οργανώσεις αλλά και στις κοπερατίβες που εμφανίστηκαν και στην περιοχή πριν κάποια χρόνια. Όμως, νομίζω ότι εμείς βρισκόμαστε εδώ για να σκεφτούμε και πώς μπορούμε να διαχειριστούμε την ε, κοινή γεωργική πολιτική για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Εγώ βλέπω εδώ ε, ότι έχουμε οργανώσεις μόνο στη, σε ό,τι αφορά τα όχι στους άλλους τομείς. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε συνολικά την κατάσταση, αλλά και στα απορροκυπευτικά βλέπουμε... Εγώ προέρχομαι από μια περιοχή όπου παράγουμε πάρα πολλά τέτοια οπροκυπευτικά και έχουμε ισχυρές οργανώσεις παραγών, όμως η συγκέντρωση στην πλευρά της διανομής είναι ακόμη μεγαλύτερη από αυτή που έχουμε εμείς. Και έχω συχνά την εντύπωση και εσείς σωστά αναφερθήκατε σε όργανα που ελέγχουν τον ανταγωνισμό ότι ενώ ελέγχουν με πολύ μεγάλη προσοχή το γεωργικό κόσμο όταν μιλάμε για τον έλεγχο της διανομής πολλές φορές αφήνουν εκεί μεγαλύτερη ελευθερία Δηλαδή επιτρέπονται κάποιες συγκεντρώσεις και δεν επιτρέπουν πλέον το παιχνίδι να γίνεται με ισότιμους κανόνες. Αυτό ίσως λοιπόν ξεπερνά τις οργανώσεις παραγωγών. Εμείς είχαμε μακρά συζήτηση για ε, τον θέμα των κοινοπραξιών, τα κονσόρσια γιατί πολλές φορές ε, έχουν μεγαλύτερες διαστάσεις από τις οργανώσεις παραγωγών. Έτσι λοιπόν, ε, εσείς ε, μπορείτε να φανταστείτε στα πλαίσια του δικαίου του ανταγωνισμού ακόμη μία πιο μεγάλη συγκέντρωση σε σχέση με αυτή που μπορεί να προσφέρει μία οργάνωση παραγωγών για να απαντήσουμε στις προκλήσεις των μεγάλων διανομέων που παίζουν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα. Πόσο Ε. φλάνακαν. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα. Όλα αυτά θέλω ιδιαίτερως ε, να εστιαστώ στις οργανώσεις παραγωγών και κυρίως επιπλέον τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με, με το ποιον συναλλάσσεται ο παραγωγός και κυρίως το μέγεθός του. Δεν ξέρω ποια είναι δική σας ε, γνώμη. Εμείς πάντω στην Ισλανδία είχαμε στην περίπτωση της Ryanair, η οποία αγόρασε μετοχές της Air Lingus και κατηγορήθηκε ότι έχει μια δεσπόσα, ή κινδυνεύει να εξασφαλίσει δεσπόσα θέση στην αγορά. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τη μάχη του Δαβίδ ε, κατά του Γολιάθ. Μπορεί κανείς να περικόψει τις διαστάσεις του Γολιάθ για να βοηθήσει να ενισχυθεί ο Δαβίδ. Όταν λοιπόν ε, βρίσκεται αντιμέτωπος με τον ε, προμηθευτή ο παραγωγός, τι συμβαίνει και τι συμβαίνει σε σχέση με τους όρους του ανταγωνισμού. Ο κύριος Άγνιο αναφέρθηκε στο θέμα αυτό από μια άλλη σκοπιά. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν ώστε να ελαχιστοποιήσουμε ή να περικόψουμε τα μεγέθη αυτών που είναι είτε η μεγάλη βιομηχανία του κρέατος, το μεγάλο σούπερ μάρκετ, η μεγάλη γαλακτοκομική μονάδα. Τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε για να περιορίσουμε το δικό τους μέγεθος, γιατί με ενδιαφέρον παρακολούθησα τα είπε η κυρία που μίλησε νωρίτερα που είπε ότι είδε ανθρώπους με τους οποίους ε, συνομίλησε που είχαν ε, ε, μικρά αυτοκίνητα, παλιά αυτοκίνητα γιατί ήταν απλή γεωργία ενώ ήταν κάποιοι οποίοι έκαναν εμπόριο σπόρων ή οτιδήποτε άλλο θα έβλεπε μάλλον στο πάρκινγκ ακριβά αυτοκίνητα. Εδώ υπάρχουν κάποιοι που έχουν και ιδιωτικό τζετ, όχι γιατί τα έκλεψαν τα λεφτά, αλλά γιατί απλώς έχουν πολλά λεφτά. Και τα λεφτά αυτά τα έχουν πάρει προέρχονται από γεωργούς, από τη δική μου την περιφέρεια, από την κοινότητα στην οποία εγώ ζω και ποτέ δεν γυρίσαν πίσω. Γιατί λοιπόν όταν έρχεται η ώρα δεν συζητάμε και την ανάγκη να περικόψουμε τα μεγέθη του Γολιάθ, να του κόψουμε τα πόδια όπως θα λέγαμε. Γιατί λοιπόν δεν υπάρχει ένας πραγματικός ανταγωνισμός και στη γεωργία. Τα σπλάχνα και την απόδοσή τους. Μου λένε ότι δεν υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός σε παραδείγματι ε, και μου λένε οι παραγωγοί ότι αν ε, δεν υποκύψουν στις πιέσεις δεν θα μπορούν καν να διαθέσουν το προϊόν τους. Αυτό δεν είναι αντίθετο με, τον, ε, με το δίκαιο του ανταγωνισμού. Βλέπω ότι το δίκαιο του ανταγωνισμού χρησιμοποιείται μόνο για να συνθλιβεί ο μικρός και όχι για να περικοπεί η ισχύ του μεγάλου. Όλες αυτές οι ωραίες νομοθεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ. Η ε, κυρία Πετήρα, αλλά παραβαίνετε το χρόνο που δικαιούσε ο καθένα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση προς την ε, καθηγήτρια Γιούχας. Ε, είπατε ότι δυστυχώς ε, η Κροατία δεν, περιλαμβάνεται στη μελέτη. Το έχω επισημάνει πολλές φορές. Είμαστε πια δύο χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μελέτε και έρευνε θα πρέπει να περιλαμβάνουν και την Κροατία επιτέλου. Αναφερθήκατε στο πρόβλημα της δημογραφικής γύρασης του πληθυσμού στην Ήπεθρο, στις ε, αγροτικές ζώνες. Υπάρχει όμως και το πρόβλημα της φτώχειας, ε, της φτώχειας ε, των ηλικιωμένων που διαμένουν στην Ήπεθρο. Στην Κροατία, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι μερικοί ηλικιωμένοι προσπαθούν να επιβεβαιώσουν με συντάξεις πείνας 50 με 70 ευρώ το μήνα. Ούτε για τα στοιχειώδη, ούτε για τις στοιχειώδεις ανάγκες τους ε, δεν αρκούν αυτά τα λεφτά. Ε, πώς είναι δυνατόν να πληρώνουν ε, λογαριασμούς, ε, ΔΕΗ, νερό, ούτε καν τα προστοζήν, γιατί για την τροφή τους δεν μπορούν να εξασφαλίσουν με τέτοιες συντάξεις πείνας οι γεωργοί. Επίσης, ε, πώς ε, οι υπόλοιπες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης λύνουν αυτό το πρόβλημα των χαμηλών συντάξεων για τους γεωργούς. Υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο μοντέλο, για παράδειγμα υπάρχει ε, μια κατώτατη εθνική σύνταξη για τους γεωργούς σε κάποιο κράτος, ώστε να μπορούν και οι γεωργοί να περνούν αξιοπρεπώς στα γυρατιά τους και έτσι να παραμείνουν και να διαφυλαχθούν οι παραδόσεις και η ζωή στην Ήπεθρο. Ευχαριστώ. Ο κύριος του. Στις ε, διαστροτικές αλλαγές. Ο Άλπερτ Ντεφ τις περιέγραψε λίγο σε μια αυτόματη διαδικασία, φυσιολογική διαδικασία που δεν μπορεί να ανατραπεί. Μπορεί για ορισμένε περιοχές ε, όπως η Βαβαρία να ισχύει αυτό. Υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και περιοχές όπου ε, δεν υπάρχει καν η δυνατότητα της αναζήτησης ενός αναλλακτικού εισοδήματος, είτε πρόκειται για μικρή δομή είτε για όχι. Δεν υπάρχει αναλλακτική, λοιπόν δεν υπάρχει δυνατότητα μεταλλαγής. Και έτσι, εάν ε, ακολουθήσουμε αυτή τη λογική, μεγαλύτερες δομές είναι πάντοτε εκ προημίου καλύτερες. γιατί μπορούν να βελτιώνονται διαρκώ Στην περίπτωση τη Γερμανία, Φερρυπίν, οι μεγάλες επιχειρήσεις της Ανατολικής Ευρώπη, της Ανατολικής Γερμανίας, ωστόσο παρακολουθώ ότι είναι πιο εξαρτημένε από τις μικρές, οι οποίες είναι και πιο διαφοροποιημένε, άρα και πιο καλές. Δεν κοιτούν μόνο ένα κλάδο παραγωγή, αλλά αναζητούν αλλακτικέ πηγέ εισοδήματο. Αυτή η πολιτική λοιπόν των ενισχύσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έπρεπε να προσανατολιστεί περισσότερο προ την διαφοροποίηση και την αναζήτηση εναλλακτικών εισοδημάτων. Δεν θα έπρεπε και η παραγωγή προσθεμένης αξίας σε σχέση με το παραγόμενο προϊόν να είναι ένα κριτήριο για την υποστήριξη από την ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική. Όταν παράγει κανεί ένα υψηλή προσθέμενη αξία προϊόν, προφανώ ε, πρέπει να ε, θεωρηθεί ω ε, πιο χρήσιμο, ω σε πιο καλή θέση. Αλλά βέβαια η απελευθέρωση έγινε με δεδομένη την παγκοσμιοποίηση. Ίσως έχουμε στοιχηματίσει το λάθος άλογο και θα έπρεπε να κοιτάξουμε την πολιτική των ενισχύσεων να την προσανατολίσουμε περισσότερο προς την εναλλακτική και όχι προς τις μεγάλες μονάδες. Ευχαριστώ.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 Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με, την, ε, με τα κανάλια μας, θα τα βρούμε όμως. Διερμηνία ε, ε, υπάρχει, δεν υπάρχει πρόβλημα, απλώς με τα κανάλια λάθος. Okay. λοιπόν, θεωρώ ότι είναι σημαντικό οι θέσει εργασίας να εξετάζονται με μεγαλύτερη προσοχή. Είμαστε σε θέση ανταγωνισμού, σε μια παγκόσμια αγορά και άρα ίσως δεν είναι σωστή η προσέγγιση και η διαφοροποίηση μέτρα ταξί μικρής και μεγάλης επιχείρησης. Έχουμε δει με τις ενισχύσεις μέχρι τώρα κεφαλαιοποίηση με βάση τις τιμές της γης αλλά αυτό δεν έχει φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και γι' αυτό νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναλύσει τους διαφορούς κανονισμούς και τις διατάξεις που ισχύουν και με στα κράτη και μεταξύ κρατών, γιατί υπάρχουν άμεσα ενισχύσεις ορισμένων κρατών, ενώ σε κάποια άλλα είναι υποχρεωμένος ο παραγωγός να διαφυλάσει και κάποιους κανόνες περιβαλλοντικούς που ανεβάζουν ασφαλώς το κόστος του. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ισχύουν ίσες συνθήκες για όλους. Και γι' αυτό τίθεται το ερώτημα εδώ, πώς μπορούμε να έχουμε ίδιους ταυτόσιμους κανόνες μεταξύ των κρατών. Και πώς οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις, μεγάλες και μικρές, μπορούν να φτάσουν στην αξιοποίηση της τελευταίας τεχνολογίας. Φερρυπίν για την ε, ε, για τον καθαρισμό των γεών από αμμονία και άλλες ε, ζημιογόνους ουσίες, πράγμα στο οποίο μπορεί να έχει προχωρήσει κάποια χώρα όπως η Γερμανία, ακόμα περισσότερο η Δανία, η οποία έχει και απαγόρευση ακόμη επιβάλλει. Γιατί ξέρουμε ότι αυτές οι μέθοδοι για τον καθαρισμό των εδαφών, η χρήση νέας τεχνολογίας, μηχανημάτων κτλ. ανεβάζουν και την τιμή. Το κόστος και άρα και την τιμή του προϊόντος. Δεν μπορούμε να έχουμε ε, τέτοια διαφοροποίηση. Και πάντως δεν χρειάζεται διαφοροποίηση μεταξύ μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων. Ο κ. Μπόκοβιτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, Όταν μιλούμε για γεωργικά μοντέλα, κατέστη σαφέ ότι υπάρχει ένα σχετισμό μεταξύ του μεγέθου τη γεωργική εκμετάλλευση και των δραστηριοτήτων που διεξάγονται σε αυτήν. Βέβαια, αυτό ο σχετισμό φαίνεται ότι όλο και ευθύνει. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι γεωργία ή διγεωργία που δημιουργούνται και σχετίζονται με την ποικιλομορφία και τη διαφοροποίηση. Και αυτή η τάση θα συνεχιστεί. Γιατί είναι πεπερασμένο αγαθό η γη. Αλλά υπάρχουν και άλλες επιλογές. Εγώ είμαι από τη Σλοβενία για παράδειγμα και μπορώ να πω ότι όλο και περισσότεροι νέοι προτιμούν ε, να ζουν στην Ήπεθρο, στη φύση, είναι υπέρ της οικολογικής γεωργίας, της βιολογικής γεωργίας, υπέρ των ε, βραχιών αλυσίδων διανομής. Αγοράζουν όποια προϊόντα υπάρχει καλύτερο συντονισμός με τις ε, κοινοφελείς υπηρεσίες, ε, βοήθεια στους ε, ε, βοήθεια στους ανθρώπους με δικές ανάγκες. Απομακρυνόμαστε από τα κλασικά μοντέλα. Έχουμε όλο και νέους τρόπους ε, ανάπτυξη γεωργική δραστηριότητας και σε αυτή τη διαφοροποίηση θα πρέπει να επενδύσουμε για να δημιουργήσουμε και νέες θέσει απασχόληση. Ευχαριστώ. Ο κύριο Άγγινιο, παρακαλώ. Ευχαριστώ για τη δεύτερη ευκαιρία που μου δίνετε. Καθώ με ανέφερε ο κύριο Φλάνεγκαλ, θα ήθελα να απαντήσω, ίσως ε, να μην εννοούμε τα δύο πράγματα. Το παράδειγμα που θα σας δώσω για το πώς δουλεύει το δίκαιο του αγωνισμού στη Βρετανία είναι το εξή. Ε, έχουμε το δύο ε, παραγωγούς που συσκεύαζαν αυγά, οι οποίοι συγχωνεύτηκαν και οι Βρετανικές αρχές είπαν δεν μπορείτε να συγχωνευτείτε είστε πολύ μεγάλοι γιατί τότε θα αυξηθεί η τιμή των αυγών για τον καταναλωτή. Έτσι λοιπόν σας διατάσσουμε να διαλύσετε τη συγχώνευση. Αυτό συνέβη. Μάλιστα. Θα δώσω το λόγο στους πυρογνώμονες μας τώρα, στο 1 τέταρτο που μας έχει απομείνει δυστυχώς, 5 λεπτά στον καθένα για να απαντήσουν στις ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών. Επίσης, θα ήθελα να σας παρακαλέσω συνολικά 15 λεπτό. Ναι, ναι, συνολικά. Ένα τέταρτο μας έχει απομείνει. Θα ήθελα λοιπόν να αγγίψετε και στις αιτίε. Ε, για τη διατήρηση της κοινής πολιτικής. Γιατί εγώ πιστεύω ότι η γεωργία μας ανα... οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις επιβιώνουν χάρη στην κοινή γεωργική πολιτική και δεν μπορούν να λειτουργήσουν διαφορετικά στο Νότο για παράδειγμα. Εκεί έχουμε ελαιόδεντρα πολλά, ελαιόλαδο σε μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ακόμη και παραγωγή ε, δημητριακών, Γεωργή δημητριακών ή για την παραγωγή χειροκρέατος ε, σε άλλες χώρες. Έχουμε περισσότερο μικρές εκμεταλλεύσεις. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια μετατροπή στο ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο ίσως. Γιατί όσο πιο κλειστό είναι το μοντέλο, τόσο λιγότερο ευάλωτο στις εξωτερικές επιρροές. Από τη στιγμή όμω που έχουμε παγκοσμιοποίηση, εντατικοποίηση τη παραγωγή, βιομηχανοποίηση τη παραγωγή. και το μοντέλο είναι η παγκόσμια κοινή αγορά, τότε και εμεί, το ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο θα πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες θα θέλει να παραμείνει ανταγωνιστικό. Θα πρέπει λοιπόν να τονίσουμε την ανάγκη ενίσχυση τη ανταγωνιστικότητα στην ΚΑΠ, τη στήριξη του γεωργικού εισοδήματο, να λάβουμε υπόψη φυσικά και το περιβάλλον και είναι σίγουρο ότι οι μικρές ε, εκμεταλλεύσεις ε, δίνουν μεγαλύτερη ασφάλεια στην κοινωνία και εμπνέουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Αλλά δεν είναι αρκετά αποδοτικέ ε, και δεν εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπέ γεωργικό εισόδημα. Θα πρέπει λοιπόν και αυτό να το λάβουμε υπόψη. Γιατί μπορεί να μιλάμε για τις ωραίε γεωργικές εκμεταλλεύσει, αλλά η πραγματικότητα για αυτέ είναι πολύ σκληρή. Και παρόλο που ε, θέλουμε και η καρδιά μας ε, βρίσκεται στις μικρές ε, εκμεταλλεύσεις, η αδύρυτη οικονομία οδηγεί προς άλλη κατεύθυνση. Θα παραμείνουν οι Γεώργοι στις μικρές εκμεταλλεύσεις, αν δεν μπορούν να επιβιώσουν. Μάλλον όχι. Παρακαλώ, θα ήθελα και αυτό να το σχολιάσετε. Thank you again, uh, Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε ότι το μέγεθος ε, δεν έχει σημασία. Δεν είναι καθοριστικό. Ας το εξετάσουμε εκ του σύνεγγες αυτό. Ναι, από τη μια πλευρά, στην πραγματικότητα ε, και στις γεωργικές δραστηριότητες, ε, όντως το μέγεθος δεν μετράει πια. Το τόνισαν και οι κύριοι Ντεκάστρο, Μπόκοβιτς, Ντόρφμαν, Χόισλινγκ. Ο κόσμος βρήκε λύση στην πράξη, στη διαφοροποίηση, στις πολλαπλές δραστηριότητες, στην ανάπτυξη ε, γεωργίας χαμηλού κόστους, στη δημιουργία νέων ευκαιριών για μεταποίηση των προϊόντων στην γεωργική εκμετάλλευση και στην αναζήτηση νέων διεξόδων στην αγορά. Οπότε ε, όντως έχουν βρεθεί λύσεις και έβεσαν ενέπτυξε 11 διαφορετικές στρατηγικές που χρησιμοποιούνται επί το, στην πράξη ώστε να δημιουργηθεί γεωργικό εισόδημα άσχετα με το μέγεθος της αγροτικής εκμετάλλευσης. Ο κόσμος έχει βρει λύσεις. Το θέμα βρίσκεται και το πρόβλημα βρίσκεται σε επίπεδο γεωργικής πολιτικής και σε επίπεδο κοινή γεωργικής πολιτικής το μέγεθος μετράει. Και έχουμε μια παράδοξη κατάσταση όπου οι άμεσε ενισχύσει πηγαίνουν στι μεγαλύτερε. Ε, φάρμες, μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις. Και σας εγγυώμαι ότι θα ασκηθούν μεγάλες πιέσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη να συνεχιστεί αυτό το σύστημα, ε, έστω και μερικώς, και μετά το 2020. Σίγουρα θα ασκηθούν ε, μεγάλες πιέσεις υπέρ της διατήρησης αυτού του συστήματος. Και στον δεύτερο πυλώνα, στην ανάπτυξη της υπαίθρου, υπάρχει ε, περιορισμός, να μην δίνονται ενισχύσεις στις ε, μικρές κυρίως επιχειρήσεις που έχουν πολλαπλές δραστηριότητες, που έχουν διαφοροποίηση. Υπάρχει λοιπόν διακριτική μεταχείριση και μεγάλη επιλογή στην κατανομή των ενισχύσεων. Εκεί θα πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές λοιπόν. Και υπάρχει και το θέμα αυτό που επισήμανε ο πρόεδρος. Πού θα πηγαίνει η ενίσχυση, στο περιβαλλοντικό σκέλος, στο ανταγωνιστικό σκέλος, στο σκέλος της παραγωγής, στην παραγωγικότητα. Εγώ θα έλεγα ότι ήδη υπάρχει η λύση στην πράξη και εφαρμόζεται. Έχουμε στην Ευρώπη τρόπους γεωργικής υποκαπιτάλευσης που είναι και ανταγωνιστική και φιλοπεριβαλλοντική και αποδοτική με υψηλή παραγωγικότητα. και μεγάλα επίπεδα παραγωγικότητας μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς ε, κατά ανάγκη ε, γεωργία μεγάλης κλίμακος. Οπότε σε αυτά τα σημεία θα πρέπει να επικεντρωθεί η νέα γεωργική πολιτική. Επίσης αναφέρθηκε αυτό το δίλημα μεταξύ των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων και των μεγάλων ε, εκμεταλλεύσεων που συγχωνεύονται στη Γεωργία. Αυτό είναι πρόβλημα όντως. Γιατί στις, στις, στην Αιθιοπία, στην Ουκρανία, στο Μαγκρέπ, στη Σενεγάλη, στην περιφέρεια της Ευρώπης ε, αναπτύσσονται μεγάλοι όμιλοι. 1.200 εκτάρια αρδεύσιμες καλλιέργειες ποροκυπευτικών ε, στο Μαρόκο σε σχέση με πολύ μικρότερες ε, εκτάσεις στην Ολλανδία. Αυτό απειλεί, αυτή η συγκέντρωση απειλεί τις μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Τέτοιου όμως μεγάλες εκμεταλλεύσεις μπορούν να εμφανιστούν και στην Ευρώπη εξαιτία της ε, αλληλεπίδρασης δύο παραγόντων. Καταρχήν, οι, οι τράπεζες είναι οι ιδιοκτήτες ε, μεγάλων μεγάλων εκτάσεων και επίσης έχουμε μη ε, γεωργούς επιχειρηματίες που έχουν για κερδοσκοπικούς λόγους να επενδύσουν τα κέρδη τους στη γεωργία. Κάτι τέτοιο ίσως ε, οδηγήσει στην ε, εμφάνιση μεγάλων αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρώπη που θα είναι ιδιαίτερα επιζήμιες στην οικογενειακή γεωργία, στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Και φυσικά δεν θα, δεν θα αναπτύξουν θεμητό ανταγωνισμό αυτές οι μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Οπότε η νέα ΚΑΠ θα πρέπει να προφυλάξει τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις αυτό το επιθετικό νέο πλαίσιο που θα δημιουργηθεί. Επίσης μελέτησα το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4 Φεβρουαρίου του 2014 με θέμα το μέλλον των μικρών ε, αγροτικών εκμεταλλεύσεων και το ψήφισμα τα λέει όλα με σαφήνεια. Τώρα όμως θα πρέπει να δοθεί σάρκα και ωστά στις προτάσεις αυτές, στις συζητήσεις για το νέο, στις νέο των συζητήσεων για τη μελλοντική εκείνη γεωργική πολιτική. Η κυρία Γιούχας. Έχω μία ερώτηση. Έχω μία ερώτηση. Εγώ ήμουν ο συντάκτης ε, αυτής της έκθεσης για τις μικρές εκμεταλλεύσεις. Και όλοι συμφωνήσαμε ως προς το περιεχόμενο όταν το συζητήσαμε. Όταν όμως χρειάστηκε να διατυπώσουμε κάποιες αλλαγές για την κοινή γεωρική πολιτική, τότε ξεχάσαμε τι είχαμε προτείνει στην έκθεση. Παρακαλώ. Well, in the first place... Ναι. Καταρχάς πρέπει να πω ότι με τιμά ιδιαίτερο το ότι κάθομαι στο τραπέζι με τον συντάκτη ενός τόσο σημαντικού ψηφίσματο. Σας ευχαριστώ πολύ και μακάρι να μπορέσω να σας βοηθήσω για να επισημανθεί για μια φορά το θέμα στο Κοινοβούλιο με πολύ εύστοχο τρόπο. Περιγράψατε τη σημασία των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων για την παραγωγή τροφής στην Ευρώπη, για το περιβάλλον, για την κατάρτιση. Και επιπλέον θα ήθελα να πω ότι πρόσφατα είδα και μια παρόμοια έκθεση της Γερουσίας των Ηνωμένων που ακολουθεί ακριβώς την ίδια επιχειρηματολογία. επισημένοντας ένα από τα ελαττώματα της Γενικής Διευθύνσης Γεωργίας ότι είναι υπερβολικά προσανατολισμένη στι ε, στις εξαγωγές και γι' αυτό επιμένει ιδιαίτερα στην ε, ανάγκη για μεγάλες και ανταγωνιστικές εκμεταλλεύσεις και δεν σκέφτεται σε όρους περιφερειακής οικονομίας και τις ανάγκες αυτής ή τις δυνατότητες μπορεί να παραχθούν σε αυτό το επίπεδο γιατί αν το κάνει κανείς αυτό βλέπει διαφορετικά την εικόνα, δεν είναι μικρές δεν είναι μικρές και μέσα σε εκμεταλλεύσεις πρόβλημα, αλλά ουσία για την Ευρώπη και ευκαιρία. Σας ευχαριστώ. Κύριε Καθηγητή, γιατί η συζήτηση μπορεί να πάει πολύ μακριά. Ευχαριστώ πολύ για τη Ρωσία. Για την Κροατία, συγγνώμη δεν είναι βέβαια θέμα να μην συμπαθούμε την Κροατία, να μην θέλουμε να την περιλάβουμε. Απλώς δεν είχαμε στατιστικά στοιχεία. Για λόγους ε, πρακτικούς. Ελπίζω την επόμενη φορά να είμαι σε θέση να την συμπεριλάβω. Για τον κύκλο υπήρξε, κάπως επελήθη το ζήτημα και πιστεύω ότι των γενναιών Νομίζω ότι τώρα, τουλάχιστον στη δική μου, στο δικό μου το κλάδο, βλέπω αλλαγή. Και γι' αυτό είναι σημαντικά τα δεδομένα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε. Σε ποιον θα ανήκουν, τι είδου πληροφορία θα αντλήσουμε και γνώση από αυτά. Πώ θα τα χρησιμοποιήσουμε για να στηρίξουμε επιλογέ, είτε σε επίπεδο γεωργία, είτε σε επίπεδο πολιτική επιλογή. Είναι και ζήτημα και νέων δεν μιλούμε μόνο για αλλαγή από τη μια γενναία στην άλλη, τόσο όσο αλλαγή τακτικής ή γενναίων. Και γι' αυτό πρέπει να προετοιμαζόμαστε. Και αν δεν προετοιμαστούμε, το χάσμα μεταξύ κεντρικής, ε, δυτικής και ανατολικής Ευρώπης θα είναι όλο και μεγαλύτερο. Και γι' αυτό εστιάστηκα το, σε αυτή τη διάσταση. για το κατά μπορεί να είναι ελκυστική η γεωργική δραστηριότητα. Βεβαίω και είναι γεγονό αυτό που είπα, γι' αυτό χρειάζεται και προαγωγή, προβολή τη γεωργική δραστηριότητα. Μπορεί να είναι εξίσου ανταγωνιστική, μοντέρνα ε, και καθαρή ε, από την λάσπη η γεωργία όσο και οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα και νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το λάβουμε υπόψη και για την προσεχή κοινή γεωργική πολιτική, γιατί πρέπει να γίνει πιο μοντέρνα η γεωργία. Για την απλούστευση. Βεβαίως, καταλήγει πάντα στο να περιπλέκει τα πράγματα. Και κάτι ακόμη, είχα την εντύπωση από τα όσα ακούστηκαν ότι ή μάλλον για τη στρατηγική. Εγώ είχα την χαρά τρεις φορές να διατυπώσω στρατηγική για, το, για την υπηρεσία θεστικής ασφάλειας, ε, στη συνέχεια για την υπηρεσία ε, γεωργικού σχεδιασμού της Ουγγαρίας και μετά ε, σε δικούς μου όρους. Και τελικά καταλήγουμε μετά την ανάλυση όλων των δεδομένων ότι ο στόχος δεν μπορεί να λύσει κάθε πρόβλημα. Αυτό είναι πάντα το πρόβλημα μια στρατηγική. Έχω την εντύπωση από τη συζήτηση ότι γίνεται μια προσπάθεια να επιληθεί κάθε πρόβλημα, μικρό και μεγάλο. Μετά όμως από κάποιο διάστημα ενασχόληση με την υπόθεση, καταλήγει κανείς βέβαια στο συμπέρασμα ότι καλό να υπάρχουν στόχοι, αλλά στην πρακτική περιορισμένες είναι οι βελτιώσεις που θα φέρουν πραγματική αλλαγή στην καθημερινή ζωή του Γεωργού η καινοτομία, η αλλαγή γενιάς, η τεχνολογία της πληροφορικής μπορούν, αλλά βέβαια και τα δεδομένα πάνω στα οποία θα στηριχθούν οι αποφάσεις μπορούν να βοηθήσουν και το τελευταίο για την φτώχεια, τη φτώχεια στην Ήπεθρο. Δεν έχω απάντηση, δεν έχω λύση. Ωστόσο αναγνωρίζω το πρόβλημα. Και το αναγνωρίζω ως τέτοιο. Διότι όσοι έχουν μείνει στις φτωχές περιοχές της υπαίθρου δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Είναι οι συνθήκες αυτές που δεν μπορούν να μετακινηθούν στα αστικά κέντρα. Δεν έχω λύση λοιπόν στο πρόβλημα. Ελπίζω η νέα κοινή γεωργική πολιτική να δώσει απαντήσεις και λύσει στο πρόβλημα. Ο Πρόεδρος ευχαριστώ πολύ. Και για, για να κατανοήσουμε τις αλλαγές και εξελίξεις στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη πρέπει κανείς ε, να έχει υπόψη ότι ε, το χωριό, η Ήπεθρος, ανήκε στα κράτος. Κατά 20% είχε την κατοχή του, του χωριού και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων το κράτος. Όλα τα υπόλοιπα ίσως, ναι. Αλλά αυτή είναι η βάση εκκίνησης. Είναι δύσκολο το πρόβλημα, όπως είπατε και εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος καθηγητής για τα τελευταία πέντε λεπτά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους για τις ερωτήσεις ε, που μου θέσατε. Δεν είναι εύκολη απάντηση. Σίγουρα τονίστηκε ένα σημαντικό θέμα ότι η οργάνωση της αγοράς είναι ένα είδος ε, μηχανισμού πρόθεσης μεταξύ μιας ε, διαρθρωτικής διαδικασίας πολύ δυναμικής ε, που είναι εκτός της γεωργίας και μίας διαδικασίας διαρθρωτικής προσαρμογής πολύ πιο βραδέως ρυθμού στη γεωργία. Και εκεί βλέπουμε ότι και μικρές μονάδες μπορούν να γίνουν ανταγωνιστικές. Όμως αυτό εξαρτάται από το πώς λειτουργεί η οργάνωση της αγοράς. Τα όσα μας είπε ο κύριος Τεκάστρο είναι διαφωτιστικά, όπως παραδείγματο χάρη μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται μόνο σε ένα μισεκτάριο μπορεί να είναι ανταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά. Αυτό χάρη σε μια οργάνωση παραγωγών που τι έκανε, έκανε μια τεράστια επένδυση στο να ταυτοποιήσει και να προωθήσει την ποιότητα ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Έκανε μια πολύ μεγάλη επένδυση στις εμπορικές υπηρεσίες και έδρασε έτσι ώστε να μπορεί να είναι ένας σημαντικός συνομιλητής πολλών αγοραστών και έτσι αύξησε και τη διαπραγματευτική του θέση. Αυτό είναι το τυπικό ευτυχές παράδειγμα, αλλά μπορούμε να εξαγάγουμε αυτό το παράδειγμα και σε άλλες πραγματικότητες, αυτό είναι το ζητούμενο. Έγινε αναφορά σε ένα σύστημα που λειτουργεί στα οπορεκπαιστικά, νομίζω, είπε ο κ. Ντόρφμαν. Όμως ε, στους άλλους ε, κλάδους ε, εξακολουθεί να έχει δυσκολίες να αναπτυχθεί. Αλλά ακόμη και στα οποροκυπευτικά συνυπάρχουν καταστάσεις όπως αυτή της επιχείρησης του Τρεντίνο με άλλες καταστάσεις όπου θεωρείται ο επιχειρηματίας ως ένας γραφειοκρατικός δεσμός παρά ως ένας παράγοντας που θα διευκολύνει την θέση σε εμπορία του προϊόντος του. Τώρα, ποια είναι τα ευτυχή μοντέλα που πρέπει να εξεγάγουμε; Σίγουρα ε, η ε, κοπερατίβα διαφέρει πάρα πολύ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά αυτό είναι ένα όριο. Υπάρχει και κάτι ακόμη όμως. Ότι έχουμε αποκλίνουσες συνθήκες. Εγώ παρέλειψα αυτή τη διαφάνεια που είχε να κάνει με υποθετικές συστάσεις πολιτικής που προσεγγίζουμε στην ανάλυση μας. Είπαμε ότι τα οποροκυτσιστευτικά υπάρχουν κάποια συστήματα, κάποιες εξαιρέσεις από τον ανταγωνισμό για το γάλα. Έχουμε ένα διαφορετικό πακέτο με διαφορετικές δεσμοί μέτρων για τα νέα προϊόντα. Τα άρθρα 169-171 του νέου κανονισμού, τις αρρώσιμες εκτάσεις ε, και τα ελαιούχα εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορετικές ε, συνθήκες και διάφορες εξαιρέσεις από τον ανταγωνισμό. Πάμε τώρα σε καταστάσεις όπου εξαιρέσεις από τον ανταγωνισμό επιβάλλουν πάρα πολύ περιοριστικούς όρους όπως στην περίπτωση του ελαιολάδου ε, και στα κρέατα παραδείγματος χάρη σε καταστάσεις ε, όπου για να μπορεί κάποιος να χέρι της εξέτασης του ανταγωνισμού είναι πολύ πιο ελαστικό το καθεστώς, όπως τα οπροκυπευτικά, παραδείγματος χάρη. Είναι προφανές ότι αυτές οι αποκλήσει μεταξύ των τομέων που πολλές φορές αιτιολογείται από πολιτικές αλλά όχι από διαρθρωτικές συνθήκες του κλάδου μπορεί να επιφέρει διαστρέβλωση των κινήτρων στους γεωργούς. Εκεί όπου υπάρχουν εξαιρέσεις ε, ε, στον ανταγωνισμό, θα μπορούσαμε να έχουμε πλεονεκτήματα για τις οργανώσεις παραγωγών, ε, ενώ έχουμε άλλους όρους σε άλλες προϋποθέσεις. Πάντοτε όμως υπάρχει ο κίνδυνος να ξαναμπίουν από το παράθυρο οι στρεβλώσεις των κινήτρων που έστειλε εκτός από την πόρτα η ΚΑΠ με την ενοποίηση των νέων πληρωμών. Έτσι λοιπόν υπάρχει αναγκαιότητα απλούστευσης και εναρμόνισης της νομοθεσίας σε ό,τι αφορά τις εξαιρέσεις των αγροτικών προϊόντων από τον ανταγωνισμό. Από το δίκαιο του Βεβαίως πρέπει να έχουμε περισσότερη ασφάλεια δικαίου Τώρα βρισκόμαστε στην εξή κατάσταση. Η Επιτροπή έχει κάνει κάποιε ερμηνευτικέ κατευθυντήριε γραμμέ αυτών των εξαιρέσεων, όμω αυτέ οι κατευθυντήριε γραμμέ αφορούν μόνο κάποιου τομεί και όχι άλλου. Και φυσικά αυτό δημιουργεί ερμηνευτική αβεβαιότητα. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που στο βαθμό που μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μία ομοιογενή εικόνα για τις εξαιρέσεις από τον ανταγωνισμό θα μπορούσαμε να υπερβούμε και έναν άλλο όρο, δηλαδή τον όρο ότι οι οργανώσεις θα πρέπει να αφορούν ένα και μόνο προϊόν, αλλά να δώσουμε τη δυνατότητα σε οργανώσεις παραγωγών να αφορούν πολλά προϊόντα, να είναι πολυκλαδικές. Αυτό για να μπορούν να κάνουν ένα σχεδιασμό και αναφέρομαι στο άρθρο 170-172 του κανονισμού 1308 αλλά θα πρέπει να τους δώσουμε και δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας στο εμπορικό επίπεδο. Όλα αυτά επιζητούν απλούστευση και εναρμόνιση. Τελειώνω. Σας ευχαριστούμε και λυπούμε που τουλάχιστον τις απαντήσεις σας χρειάστηκε να σας τις περιορίσω σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα αλλά πραγματικά επεκταθήκαμε πολύ στη συζήτηση ακριβώς επειδή ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και οι δικές σας ομίλειες αλλά έχουμε και άλλα θέματα και γι' αυτό θα πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτό το τμήμα τη συνεδρίαση για να περάσουμε στα επόμενα. Πάντω, θεωρώ ότι αυτό το σεμινάριο εμπλούτησε πολύ τι γνώσει μα και τη συζήτηση και θα αξιοποιήσουμε όλες αυτές τις γνώσεις που μας μεταφέρατε στις δραστηριότητές μας. πάμε που χρειάστηκε να σας ε, αναγκάσω να μιλήσετε πολύ πιο λίγο και να σας περικόψω το χρόνο. Σας ευχαριστούμε θερμά. Πέναμε στο σημείο 4 τη στρατηγική για τις Άλπες, για την περιοχή, την περιφέρεια των Αλπών. Η αρμόδια κατ' ουσίαν ε, για το θέμα αυτό επιτροπή είναι η Επιτροπή Ανάπτυξης, Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, που θα συντάξει έκθεση πρωτοβουλίας. Εμείς αποφασίσαμε να συντάξουμε γνωμοδότηση. Συντάκτριά μας ε, είναι η κυρία Ουλρικέ Μίλλερ, στην οποία δίνω και το λόγο. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τη γνωμοδότηση της Επιτροπής μας για τις, για τις Άλπες. Δυστυχώς ε, είμαστε υποχρεωμένοι να περιοριστούμε ως προς, τον, ε, ως προς την έκταση του κειμένου, ως προς τους χαρακτήρες δηλαδή που θα έχει αυτή η γνωμοδότηση. Ελπίζω να μπορέσουν να με βοηθήσουν και οι συνάδελφοι ώστε να κάνουμε με τις τροπολογίες ε, συμπληρώσει σε κάποια σημαντικά ζητήματα. Θέλω καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη στρατηγική, για την ε, για το χώρο των Αλπαίων για την ενασχόληση με αυτή τη στρατηγική. Το πρόγραμμα δράσης μέχρι τώρα υπάρχει μόνο στα αγγλικά, από ό,τι γνωρίζω, αλλά θα θέλαμε να το είχαμε στα, στις τρεις ε, γλώσσες εργασίας, δεδομένου ότι αφορά τις Άλπης. Και ιδιαίτερα θέλουμε να καλωσορίσουμε τη στρατηγική αυτή διότι υπογραμμίζει και τη σημασία του χώρου αυτού ως χώρου ζωής, διαβίωσης δηλαδή, αλλά και αναψυχής του χώρου των Άλπαιων και την ανάγκη για διαφύλαξή του, κάτι το οποίο χωρίς ε, λειτουργούσα γεωργική οικονομία ε, και δάσο κομία δεν μπορεί να διατηρηθεί και να προσφέρει τη συμβολή του σε ένα υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικό, παραγωγής τροφίμων, αλλά βέβαια και διαβίωσης. Όπως επίσης ε, είναι απαραίτητη και η διαφύλαξη και των παραδόσεων διαβίωσης και των οικοσυστημάτων. 48 είναι οι περιφέρειες, 7 τα κράτη και έχουμε καταγράψει 9 σημεία, εκείνα τα οποία θεωρούμε καταρχάς πολύ σημαντικά την ε, ε, ε, εγκατάλειψη από τους μόνιμους κατοίκους εν γέννη, την φυγή από την Ήπεθρο γενικότερα, την εγκατάλειψη του τοπίου αυτού και την ανάγκη για να διαφυλαχθεί το τοπίο και οι παραδόσεις του με την γεωργία κυρίως και τη δασοκομεία, εάν συνεχιστεί δηλαδή αξιοποίηση της γης και των δασών. Εδώ έχουμε να κάνουμε και με τη διαφύλαξη των ειδών, της βιοπικιλότητας, ε, των υδάτινων πόρων και ούτω καθεξής. Ένα άλλο σημείο σημαντικό είναι αυτό που έχει να κάνει με την κυριότητα και την έγκυο ιδιοκτησία και την προστασία των ε, οικογενειών των γεωργών. Περιγράφουμε αυτό που πρέπει να διαφυλαχθεί ε, με παραπομπές και στην οδηγία για το έτοιμα και για την κλωρίδα και πανίδα επίσης ε, γεωργικές δομές που περιγράφουμε και λέμε ότι η παραδοσιακή γεωργική εκμετάλλευση και κτηνοτροφία πρέπει να διαφυλαχθούν στις ορεινές περιοχές και να γίνει εναρμόνιση των εθνικών πλαισίων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση η μείωση των διδικασιών ελέγχων και της διασταυρούμενης συμμόρφωσης έχει πολύ μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα για τις ορεινές ε, περιοχές. Πέμπτον, καταγράφουμε την, ε, τις δομές διαχείρισης και διάθεση στην αγορά των προϊόντων που θα πρέπει να γίνουν με πιο στοχευμένο τρόπο, με οργανώσεις παραγωγών, συνεταιρισμούς, λέμε ότι θέλουμε μια πιο εμφανή θέση και λειτουργία, δράση καλύτερα μέσα στην αλυσίδα διάθεση των προϊόντων. Ε, αναφερόμαστε στην απασχόληση, στην καινοτομία, στις περιοχές, παραδείγματι έχουμε κοινότητες δασοκομικής δραστηριότητας με πολύ μεγάλη σημασία και για την παροχή συμβουλών πλέον δεν προσφέρει το κράτος στη Γερμανία και, γενικά, και ειδικότερα τη Βαβαρία. Ε, και επίσης η καινοτομία, η έρευνα, τα κέντρα καινοτομίας. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την ανάγκη να ενισχυθούν συγκεκριμένα, στοχευμένα, γιατί ιδιαίτερα προς την ε, φύλαξη και αξιοποίηση του ε, πρασίνου, του υπαίθρου, την κτηνοτροφία χρειαζόμαστε την υποστήριξη των ερευνητικών κέντρων. Ιδιαίτερα σημαντικό για μένα είναι να γίνεται η έρευνα ε, με στόχο τη μεταφορά στην πραγματική δράση, στην γεωργία, με απτά δηλαδή αποτελέσματα, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει πάντοτε, οι παραδοσιακές μορφές εκμετάλλευσης γεωργικής και εκτινοτροφίας μπορούν να διαφυλαχθούν μόνο χάρη στην μέθοδο των βέλτιστων πρακτικών, με την έρευνα βέβαια και την καινοτομία παράλληλα. Στο σημείο 7 αναφερόμαστε στην πρόσβαση μιας καλύτερης κατάστασης, μιας ευρύτερης επιμόρφωσης. Και εδώ, μια και είναι μικρές ε, πολλές φορές οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις ορεινές περιοχές και της Άλπης, χρειαζόμαστε ε, να παρέχονται από ειδικού οι συμβουλευτικές υπηρεσίες. παραδείγμα, υπάρχει γεωργική ακαδημία όπου ο γεωργός πέραν της επαγγελματική του δραστηριότητας έχει και 700 ώρες 720 ώρες μαθήματος, χάρη στις οποίες παίρνει και το σχετικό δίπλωμα, την πιστοποίηση ότι μπορεί να εκμεταλλεύεται την γη του και να κερδίζει χρήμα από αυτήν. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση στις, όταν πρόκειται για επιχειρήσεις των ορεινών περιοχών. Έχουμε πει ότι θα υπάρχουν επιπλέον ενισχύσεις ή νέα ταμεία ενισχύσει. Ωστόσο πιστεύω ότι χρειάζεται να συζητήσουμε ταχύτατα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι εναλλακτικέ δυνατότητε μπορεί να υπάρχουν. Ακόμα δεν έχω λάβει δηλαδή σαφή απάντηση για το εάν υπάρχουν αυτέ οι δυνατότητε και αν αναζητούνται στη σωστή κατεύθυνση, γιατί υπάρχουν ακόμα προβλήματα και αντιφάσει στα προγράμματα ενίσχυση. Υπάρχει επίση το πρόγραμμα Interreg, όπου μπορεί και η περιφέρεια και ε, σε πιο μικρό επίπεδο μια κοινότητα να διεκδικήσει κονδύλια και για τη γεωργία, τη γεωργική δραστηριότητα και τη δασοκομική δραστηριότητα για να τα διαθέσει στις αντίστοιχες επιχειρήσεις ε, για τη δικτύωσή τους. Γεωργία λοιπόν, δασοκομεία, τουρισμός, ε, χειροτεχνία. Όλα αυτά μπορούν βελτιστοποιημένα μέσα σε ένα κοινό κορβανά να υποστηριχθούν σε επίπεδο περιφέρειας. Νέα προγράμματα λοιπόν δεν χρειάζονται, πρέπει όμως να βρούμε λύσεις και πρέπει να εργαστούμε εντατικά για να βρούμε λύσεις με τα εφιστάμενα. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο λοιπόν και αυτή ήταν μια πρώτη επισκόπηση των εννέα σημείων με τις ε, τροπολογίες που περιμένουμε έως τις 18 Μαρτίου. Πιστεύω ότι θα έχω και την υποστήριξη και των σχεδόν εισηγητών. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά κυρία Μίλλερ. Εξαιρετική η παρουσίασή σας. Παρακαλώ οι ομιλητές να είναι σύντομοι. Χρόνο ο κύριος Ντόρφμαν. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω να προσθέσω πολλά. Διότι πιστεύω ότι η κυρία Μίλλερ έκανε μια πολύ πλήρη ε, γνωμοδότηση. Ένα-δύο σημεία μόνο θέλω να θίξω. Ε, πιστεύω ότι η γεωργία δεν μπορεί να περιγραφεί ως ε, μονοδιάστατη κατάσταση στον χώρο των Άλπαιων. Υπάρχουν περιοχές με, με παλόμενη γεωργική δραστηριότητα, ενώ κάποιες άλλες και μάλιστα πολύ κοντά σε αυτές τις επιτυχημένες περιοχές έχουν δει να τελματώνει και να, εκμεταλ... να εγκαταλείπεται τελείως η γεωργική δραστηριότητα. Έχουμε πολύ διαφορετικές λοιπόν συνθήκες, διαφορετικές προληπτικά μέτρα θα χρειαστούν ως εκ τούτου. Κοινό σε πολλές περιφέρειες και παντού στον χώρο των Άλπιων είναι η αναζήτηση εναλλακτικών παραγωγής. Έχουμε μεγάλο ποσοστό βοσκοτόπων που μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο εάν υπάρχει κτηνοτροφική δραστηριότητα και άρα και παραγωγή γάλακτος. Στη φάση στην οποία βρισκόμαστε λοιπόν θα πρέπει να επιλέξουμε εάν μπορούμε με απελευθερωμένη την, την αγορά γάλακτος να εξασφαλίσουμε διατήρηση της παραγωγής αυτής και στην της Σε ορεινέ περιοχέ λοιπόν και ιδιαίτερα στι Άλπε μπορεί κανεί να έχει την αντίποση ότι υπάρχουν μόνο μικρέ εκμεταλλεύσει που μπορούν να εξυπηρετήσουν μόνο τι τοπικέ αγορέ με τα προϊόντα του Βεβαίως είναι πολύτιμες και αυτές οι μικρές εκμεταλλεύσεις και ακούσαμε ήδη πολλές ε, παρεμβάσεις σήμερα για αυτές, αλλά ταυτόχρονα απευθύνονται σε μία αγορά και μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να συμμετέχουν ακόμα και σε μεγαλύτερων διαστάσεων αγορές και πρέπει και αυτό να το υποστηρίξουμε. Ένα άλλο πρόβλημα σοβαρό σε μεγάλο τμήμα των ε, ε, τη ζώνη των Άλπων, κυρίως της νότια Άλπης, στην Ιταλία και τη Γαλλία ειδικότερα, είναι ο κατακαιρματισμό της εγγύου Ιδιοκτησία, και γι' αυτό νομίζω ότι θα ήταν καλό να κοιτάξουμε, να βρούμε εναλλακτικέ απλουστευμένε μεθόδους ώστε να βοηθήσουμε και τον νεαρό γεωργό, ο οποίο δεν έχει μέχρι τώρα καμιά ευκαιρία να αναλάβει ε, ε, γεωργική δραστηριότητα, δεδομένου ότι είναι τόσο μικρά μικρή κλήρη και είναι πολύ δύσκολο να ε, εξασφαλίσει κανείς μεγέθη ικανά για μια γεωργική ε, εκμετάλλευση. Η πολυλειτουργικότητα που ανέφερε η συνάδελφος μας με τον τουρισμό και άλλα προγράμματα όπως το LEADER, το πρόγραμμα για την ανάπτυξη πέθρου του ίντερνετ και άλλα τέτοια μπορούν να βοηθήσουν ιδιαίτερα. Και τελευταία παρατήρηση, συχνά παραβλέπουμε την υδρογεολογική σημασία των Άλπαιων για, τις ε, γειτονικές, ε, για τα γειτονικά αστικά κέντρα. Ε, είδαμε και βέβαια τις συνέπειες στην νοτίως των Άλπιων. Έχουμε δει ότι ύστερα από σοβαρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες οι συνέπειες είναι ορατές και στην ευρύτερη περιφέρεια. Πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε κάτι για την υδρογεωλογική ρύθμιση του περιβάλλοντος αυτού ώστε να αποφεύγουμε τις υπερχιλήσεις ποταμών όπως είναι ο Πάδος, όπως είναι ο Δούναβης. Γενικά ε, μπορεί να καταγγέλει κανείς τις κλιματικές αλλαγές για, τις, ε, ε, για τα φαινόμενα αυτά, αλλά μπορούμε ασφαλώς να συγκρατήσουμε τα προβλήματα των υπερχιλήσεων, γιατί διαφορετικά οι κάτοικοι θα εγκαταλείπουν την περιοχή των Άλπαιων και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και για τις μεγαλύτερες πόλεις νοτιώς των Άλπων. Ευχαριστώ. Ωραία μας τα είπατε, αλλά μακρηγορήσατε δυστυχώς. Θα είμαι πολύ σύντομος, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Ως κοιόδης εισηγητής, εκτίμησα τη δομή της εκθεσής της και ευχαριστώ θα συνεισφέρουμε. Τώρα στα επιχειρήματα του κυρίου Ντόρφμαν θα ήθελα μόνο να προσθέσω το εξή, με το οποίο συμφωνώ ευρέω. Δεν είναι ταυτόσιμε σε όλες οι ορεινέ περιοχές, ούτε όλες οι λύσεις είναι κατάλληλες για κάθε φυσική περιοχή. Το μόνο στοιχείο που θα προσέθετα, στο είπε ο Ντόρφαν, είναι το θέμα της διαφοροποίησης. Εμείς ε, με τις γεωγραφικές ενδείξεις το κάναμε και είχαμε ενδιαφέροντα αποτελέσματα πρέπει να δούμε όπου είναι δυνατόν πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε κάποια στοιχεία διακριτότητας. Δηλαδή να μπορούν να αναγνωρίζουν μια πρόσθετη αξία καταναλωτές στα προϊόντα από τις ορεινές περιοχές και πώς μπορούμε να προωθήσουμε αυτά τα στοιχεία τα διακριτικά έτσι ώστε να δώσουμε μια προσθεμένη αξία σε αυτό το προϊόν είναι μια επιπλέον σκέψη που θα μπορούσε να εμπλουτίσει την εξαιρετική δουλειά της κυρίας Μίλλερ. <clears throat> Äh, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και εμείς είμαστε υπέρ της γνωμοδότησης. Είναι πολύ αξιόλογη η γνωμοδότηση της κυρίας Μίλλερ. Και είναι σημαντικό να έχουμε μια ειδική στρατηγική για τις ε, περιφέρειες αυτές που αντιμετωπίζουν παρόμοιες ε, προκλήσεις και θέλουν να εξασφαλίσουν βιωσιμότητα των πόρων τους χωρίς να παραμελούν και την ανάπτυξή τους. Η στρατηγική για την περιοχή των Αλπών θα μπορούσε να συγκριθεί με τη στρατηγική για τη Βαλτική, για το Δούναβι για παράδειγμα. Πάντως, ε, τα 80 εκατομμύρια ανθρώπων που διαμένουν σε ορεινές περιοχές να μην μείνουν εγκαταλελειμμένοι. Θα πρέπει κάτι να κάνουμε και για αυτούς. Βέβαια, έχουμε και το Λιχνιστάν και την Ελβετία και θα πρέπει να συντονιστούμε με τις χώρες αυτές που επίσης βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των Αλπών και στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής να έχουμε καλύτερο συντονισμό και των κονδυλίων για την περιοχή αυτή έχουμε να αντιμετωπίσουμε κοινέ προκλήσει. Τις περιγράψαμε και στο παρελθόν, να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να βελτιώσουμε την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και στη γεωργία και στη δοσοκομεία. Αλλά στο μέλλον άλλα σημαντικά στοιχεία θα είναι και το νερό, η διαχείριση του ύδατος και η ενέργεια. Όλα αυτά αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τα κλιματικά ζητήματα επίσης θα πρέπει να είναι εγκάσια και να λαμβάνονται υπόψη σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα. Να μην ξεχνούμε ταυτόχρονα και τον τουρισμό για να προσελκύσουμε περισσότερους τουρίστες ε, στην περιοχή αυτή προσφέροντάς τους ε, ποιοτικά προϊόντα. Επίσης, μεταφορές, άλλο σημαντικός κλάδος που δεν θα πρέπει να παραμεληθεί. Φυσικά, καλό θα ήταν να μην χρησιμοποιηθούν, να μην χρειαστούν νέα κονδύλια, αλλά να γίνει καλύτερο συντονισμό των υφισταμένων πόρων και κονδύλιων. Επίσης, ε, για τον τουρισμό βλέπουμε ότι έχουμε μεγαλύτερη καινοτομία, ντόπια τυριά, γεωργικά προϊόντα, φρούτα. Καλό θα ήταν όμως να έχουμε προϊόντα που να παράγονται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και όχι μόνο εποχιακά. Πάντως, επαναλαμβάνω πολύ αξιόλογη γνώματα τη κυρίας Μίλλερ. Ευχαριστώ. Δεν επέβαλα περιορισμό στις παρεμβάσεις, αλλά σας θέρμο παρακαλώ, σας οικετεύω ε, να αυτοπεριοριστείτε, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Κυρία Τέρας. Ευχαριστώ. Λέει κυρία Τόρες, θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το έργο της, γιατί βλέπω ότι έκανε εξωθαύμαστη προσπάθεια για να βελτιώσει την πρόταση της Κομισιόν. Παρ' όλα αυτά θέλω να αναφέρω κάποια σημεία. Όπως ξέρετε, πάνω από το ίμιση του ευρωπαϊκού πληθυσμού ζει σε αγροτικές περιοχές. Αυτό σημαίνει πάνω από το 21% το 91% συγγνώμη, της έκτασης, της επικράτειας. Γι' αυτό θα πρέπει να προστατεύσουμε τον τρόπο ζωής των ανθρώπων στις ορεινές περιοχές, αλλά και σε άλλες αγροτικές περιοχές, όπως και στην περιοχή των Άλπαιων, αλλά στα Πυρηναία, στα Κατάμπρια στην Ορόσυρα, στην Καντάμπρια και γι' αυτό νομίζω ότι αυτές οι στρατηγικές θα πρέπει να προστατεύουν ένα βιώσιμο τρόπο παραγωγής. Αυτό δεν είδα να αναφέρεται σε κανένα σημείο της έκθεσης. Κάτι άλλο που θέλω να τονίσω είναι ότι ακόμη και αν γίνεται στην ενίσχυση των ρόλων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, δεν βλέπω καμία αναφορά στα μικρά κυκλώματα εμπορίας. Και εγώ νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό, αν κατανοούμε την ανάπτυξη της ε, υπαίθρου ως ε, ένα σημαντικό τμήμα της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και της ενίσχυσης των τοπικών κοινοτήτων. Τέλος, θα ήθελα να δηλώσω τη δυσαρεσκιά μου γιατί στο τρίτο σημείο η σύτρία αναφέρεται ε, στην ε, ιδιοκτησία της γης και την ε, θέτει ως προϋπόθεση πάνω από τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων. Εμείς ε, εδώ δεν είμαστε εδώ απλώς για να κατακτήσουμε και να ιδιοποιούμαστε αυτό τον πλανήτη. Εμείς ε, δεν είμαστε πάνω από τον πλανήτη, απλώς ζούμε σε αυτό τον πλανήτη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για ένα λεπτό παρακαλώ κύριε Μποκόβιτς. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ την Ουλουρικέ για την γνωμοδότηση αυτή που έχει να κάνει με την περιοχή των Αλπέων. Μιλάμε για μια καλά αναπτυγμένη περιοχή στην Ευρώπη. Έχουμε πολλές ε, καλές πρακτικές σε αυτή την περιοχή και θα μπορούσαν ε, να εφαρμοστούν και σε άλλες ορεινές περιοχές στην Ευρώπη. Εδώ επικεντρώμαστε κυρίως στη Γεωργία και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσουμε τη συνεργασία και τη συνύπαρξη του περιβάλλοντος, του τουρισμού και της γεωργίας. Νομίζω ότι πολύ συχνά μιλάμε για το πώς το ένα στοιχείο αποκλεί το άλλο. Νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο πώς μπορούμε να συνεργαστούμε και να συνεπάρχουμε. Πρέπει να διατηρήσουμε την οικονομική δραστηριότητα αλλά και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όσοι θέλουν να προστατεύσουν το περιβάλλον δεν μπορούν να το κάνουν αυτό δίχως στη γεωργία και φυσικά θα πρέπει να αξιολογούμε περισσότερο και το θέμα της οικολογίας Αρμόδια κατοσύνη η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. απλώ σε γνωμοδότη συντάσσουμε. Ο κύριο Μπούντα, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε δύο κυρία σημεία. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια Νομίζω ότι σε, αυτούς, ε, σε αυτές τις περιοχές ε, έχουμε τρόφιμα υψηλής ποιότητας και χρειάζονται οι Ευρωπαίοι καταναλωτές αυτά τα προϊόντα υψηλής ποιότητας, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το πώς θα προλάβουμε την εγκατάλειψη των γεών σε αυτές τις περιοχές. Γιατί οι άνθρωποι εγκαταλείπουν αυτές τις περιοχές και αυτό οδηγεί σε περιβαλλοντικά προβλήματα. Πώς ε, θα καταστήσουμε ελκυστικές αυτές τις περιοχές μόνο μέσω της εμπλοκής των τοπικών αρχών και της δημιουργίας ε, υποδομών, κοινωνικών υποδομών όπως νοσοκομεία και σχολεία, δρόμο. Έτσι λοιπόν ε, να μπορούν να είναι προσβάσιμες αυτές οι περιοχές στο κοινό. Διαφορετικά δεν μπορείς να καταστήσεις ελκυστική μια περιοχή. Σας ευχαριστώ. Ο Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την ε, εισηγήτρια με την οποία συμφωνώ σε διάφορα σημεία της εκθεσής της. Εγώ εντάχει θα επικεντρωθώ πολύ συχνά η αγροτική παραγωγή αυτών ε, των περιοχών ε, είναι ποιοτική. Όμως δυστυχώς ε, παραμένει σε μια πολύ περιορισμένη αγορά. Ο στόχος είναι να διευρύνουμε αυτή την αγορά και μπορούμε να το κάνουμε δημιουργώντας ένα σύστημα με τους τοπικούς κλάδους όπως ο τουρισμός και η βιοτεχνία. Και μπορούμε να δημιουργήσουμε λοιπόν ένα τέτοιο ισχυρό δίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να προσδώσουμε αξία στο προϊόν και να πράξουμε έτσι ώστε να διευρυνθεί και η αγορά για τους παραγωγούς αυτούς. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ροπέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι η γνωμοδότηση είναι αρκετά καλή γιατί επισημαίνει τις ανάγκες της περιοχής των Άλπων ε, ιδιαίτερα στη Γεωργία γιατί η Γεωργία είναι πολύ σημαντική και για την περιοχή των Άλπων είναι αδιανόητη η περιοχή αυτή χωρίς το τομέα της γεωργίας. Δυστυχώς έχουμε εκτεταμένο φαινόμενο εγκατάλειψης γεών με άνθηση της άναρχης βλάστησης. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τους γεωργούς για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα στην περιοχή αυτή. Γιατί είναι μια περιοχή που μπορεί να παράγει υψηλής ποιότητας προϊόντα και αυτό και χρειαζόμαστε περισσότερο εργατικό δυναμικό. Και παρόλα αυτά και η περιοχή αυτή αντιμετωπίζει προβλήματα απασχόληση, ανεργία. Και φυσικά να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα όχι μόνο τη γεωργία, αλλά ιδιαίτερα των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Ευχαριστώ. κύριο Δημήτρου, παρακαλώ, αν μπορείτε να είστε λακωνικό, γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχά να καλωσορίσω τη γνωμοδότηση με τις προτάσεις που αφορούν και συνοριακές πτυχές για το χώρο των Άλπαιων. Η στρατηγική για τις Άλπες, όπως και άλλες μακροπεριφερειακές στρατηγικές Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στηρίζονται στην ανάπτυξη μιας περιφερειακής προσέγγισης και στοχεύουν στη βελτίωση της ισχύουσα νομοθεσίας πολιτικής ταμείων, κονδυλίων, Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, παραδείγματι και Η εφαρμογή έχει αρχίσει Τώρα έχει έρθει η ώρα να δείξουμε ηγητική στάση αλλά και να ε, ενστερνιστούμε τα ζητήματα αυτών των περιοχών του των Άλπαιων για να φέρει αποτελέσματα η στρατηγική. Ε, συνεργάζεται λοιπόν με τις ε, αρχές διαχείρισης των κρατών μελών, για τον προσδοσμό των στόχων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τις εταιρικές συνεταιριστικές σχέσεις για την περίοδο 2014-2020 βλέπουμε ένα μεγάλο δυναμικό ανάπτυξη τη ε, περιοχή και για λόγους κοινωνικού, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς νομίζουμε ότι μπορεί να αρθεί σε των προκλήσεων. Το ΦΟΚΑ, κομμάτι άλλωστε της κοινωνικής πολιτικής, είναι ένα μόνο ταμείο το οποίο μπορεί να παρέμβει στην ε, κατεύθυνση αυτή η κοινή γεωργική πολιτική προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων για να συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής της, ε, των Άλπαιων, η ανάπτυξη της υπαίθρου, όπου, όπου έχουν εντοπίσει είτε το κράτη είτε οι περιφέρειες ανάγκες ε, μπορεί χάρη στο, στη διοχέτευση, στην καθοδήγηση αυτής της στρατηγικής και των μέσων της να βοηθήσει την ελοπίση των στόχων. Καλωσορίζουμε λοιπόν τις προτάσεις και τις συστάσεις της κυρίας Μίλλερ και θεωρώ ότι επισημαίνει μια από τις πιο σημαντικές προκλήσεις του χώρο της πέτρου της Άλπης. Επιτρέψτε μου να επισημάνω κάποια από τα εργαλεία που έχουμε στην πολιτική για την ανάπτυξη της υπαίθρου για να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και πιστεύω ότι όλοι μας πρέπει να κινητοποιηθούμε περισσότερο και να, να συντονίσουμε καλύτερα τις προσεγγίσεις μας για να επιτύχουμε αυτή τη στρατηγική. Σε σχέση με την εγκατάλειψη της γεωργικής γης, ε, βιοπικιλότητα, ε, οικολογική αξιοποίηση της γης, η ενισχύσεις στους ε, γεωργούς και για περιοχές δασόδης έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη διαφύλαξη της γεωργικής δραστηριότητας δραστηριότητα και έμεσα βοηθάει και στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος αλλά και στη διατήρηση της εργασία στην περιοχή. Τα μέτρα ανάπτυξης της υπαίθρου που υποστηρίζουν την προστασία της βιοποικιλότητας όπως το Μετρό 2000 αλλά και άλλα μέτρα παρέμβαση για γεωργικές, κλιματικές αλλαγές, ε, και άλλα μπορούν να βοηθήσουν να φέρουν πλεονεκτήματα για το περιβάλλον και ταυτόχρονα να επιτρέψουν τη διαφύλαξη και ανάπτυξη νέων θέσεων εργασία και την αηφορό ανάπτυξη στην περιοχή. Με, τη γεωργική, με την ανάπτυξη της πέθρου μπορούν να καλυφθούν και πολλά ζητήματα του δασοκομικού τομέα, πολύ σημαντικού για τις Άλπεις. Αυτό χάρη είτε στη διατήρηση των δασών είτε σε γεωργικές υπηρεσίες σημαίνει ότι μπορούν να προσθέσουν, να φέρουν προσθεμένη αξία για να επιτρέψουν και την ανάπτυξη και την ε, βιωσιμότητα των δασών. Ένα άλλο ζήτημα είναι αυτό που έχει να κάνει με την ε, κατεργασία και διάθεση στην αγορά των γεωργικών προϊόντων της περιοχής και ταυτόχρονα ενίσχυση και του ρόλου του παραγωγού στην, αξία της, ε, στην αλυσίδα της αξίας και την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων. Επενδύσεις μπορούν να ε, χρηματοδοτηθούν και χάρη στα προγράμματα για την ανάπτυξη πέθρου που και λαμβάνουν έτσι υπόψη διάφορες διαστάσεις όπως ορεινές περιοχές, ε, Άλπης και το καθεξής. Μπορούμε επίση να υποστηρίξουμε το Γεωργό ενισχύοντα τη θέση του στην αλυσίδα αξιών, βοηθώντας τον να οργανωθεί σε οργανώσεις, ομάδες παραγωγών, ε, συνεταιρισμού και άλλες δραστηριότητε βέβαια μπορεί να προσφέρονται σε σχέση με την καινοτομία, την ευρωπαϊκή εταιρική σχέση για την καινοτομία, όπου μπορούν διάφορε ομάδε ενδιαφερομένων να συνεργάζονται για να εντοπίζουν τα προβλήματα και να βρίσκουν τι καταλληλότερε λύσει. Συμφωνώ ότι οι υπηρεσίε κατάρτιση παροχή συμβουλών έχουν πολύ μεγάλη σημασία και έχουμε διευρύνει το πεδίο εφαρμογή και ταυτόχρονα και τον αριθμό των δικαιούχων ε, μονομένη γεωργή, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις κτλ. Όλα αυτά λοιπόν συμπληρωματικά και με άλλα παρεμβατικά ταμεία και επίσης η διαπεριφερειακή διάσταση τελευταίο σημείο και η υπερσυνοριακή συνεργασία. Στην τωρινή πολιτική για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών έχουμε δυνατότητες να βοηθήσουμε προσφέροντας υποστήριξη σε φορείς παραγόντες μιας περιοχής, μιας περιφέρειας, διαπεριφερειακά και υπερσυνοριακά με στόχο την υποστήριξη δραστηριοτήτων που έγινε εκτός του χώρου ακόμα της συγκεκριμένη περιοχής και αυτές μπορούμε να τις υποστηρίξουμε δηλαδή. Και εν τέλει θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι έχουμε μια συνδιαχείριση με τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες. Την υπόθεση αυτή τις βοηθούμε τις ε, περιφέρειες και τα κράτη για να βελτιωθεί το πρόγραμμα. Αλλά μια και μιλούμε για συνένωση αυτών των μέσων, θα ήθελα να σας πληρώσω ότι υπάρχει μια πρόταση για συγκεκριμένα μέτρα που θα αφορούν μόνο ορεινές περιοχές. Δυστυχώ όμως υποχρεωμένο να σας ενημερώσω ότι δεν υπάρχει ακόμα αυτή η δυνατότητα. Σα ευχαριστώ πολύ. Ήδη έχουμε αρχίσει να ασχολούμαστε με το θέμα αυτό και θα συνεργαστούμε και με τα κρατημέλη και την περιοχή των Άλπαιων ώστε να βελτιωθεί η στρατηγική και να φέρει αποτελέσματα. Μάλιστα. Πολύ πλούσια συζήτηση ενδιαφέρουσα. Παρακαλώ η συντάκτρια μας αν θέλει, πολύ σύντομα όμως. Δεν χρειάζεται. Ωραία. Μέχρι τις 18 Μαρτίου έχετε δύο ώρια για τις τροπολογίες. Φαντάζομαι θα αξιοποιήσει το περιεχόμενο της συζήτησης η συντάκτηρια γραμματότης. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την καρποφόρα αυτή συζήτηση. Χωρίς άλλη χρονοτριβή περνάμε στο σημείο 5, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ για τις δόλες πρακτικές ε, στην εμπορία του μελιού. Θα δώσω αμέσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Φιλίπ Λόπερτ. Παρακαλώ. Good evening. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Φιλιπλοπίτ και είμαι επικεφαλής ε, της μονάδας ε, της χνηλασιμότητας ε, Θα θέλουμε να κάνουμε αυτή την προφορική παρουσίαση για τις ε, πρακτικές νοθείας στην εμπορία του μελιού. Σας ευχαριστώ για την ανταλλαγή απόψεων και την ε, πρόσκλησή σας. Καταρχήν το μέλι είναι φυσική ουσία που παράγεται από τις μέλισσες ε, και δεν θα πρέπει να υπάρχουν προσθήκες σε αυτό. Δηλαδή δεν θα πρέπει να έχουμε αρώματα ούτε προσθήκες ζάχαρης η τιμή ποικίλει ανάλογα με τη βοτανική πηγή του μελιού και άλλες παραμέτρους ποιότητας όπως η οργανική παραγωγή, η προέλευση κτλ. Και αυτές οι παράμετροι δεν ε, μπορούν πάντοτε να μετρηθούν ε, ή δεν είναι ορατές χωρίς ε, πολύπλοκη ανάλυση. Και αυτό δίνει τη δυνατότητα σε πρακτικές νοθείας για να αυξηθεί το κέρδος. Έχουμε τρία είδη προβλημάτων με το μέλι. Καταρχήν η νοθεία του μελιού γίνεται κυρίως με την αντικατάσταση της ζάχαρης με τεχνητή ζάχαρη. Το άλλο θέμα αφορά την λασασμένη δήλωση της βιτανικής προέλευσης και επίσης έχουμε ε, και παραποίηση της γεωγραφικής προέλευσης. Έτσι λοιπόν θα αναφερθούμε λίγο παραπάνω στο θέμα της νόθευσης, γιατί η νόθευση προκύπτει από την ε, προσθήκη ουσιών όπως νερό ή ζάχαρη. Πολύ συχνά ε, προσθέτουν ε, κάποια γλυκαντικά που προέρχονται από το ρύζι ή από το καλαμπόκι. έχουμε μεγάλες δυσκολίες να αντιμετωπίσουμε αυτές τις πρόσθετες ζάχαρες. Το μέλι είναι ένα πολύπλοκο μείγμα από φυσικά ζάχαρα. Μπορούμε να έχουμε 10 διαφορετικές ζάχαρα που αναμειγνύονται μαζί ανάλογα με την προέλευση του μελιού την βοτανική του προέλευση και επομένως είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε μια πρότυπη σύνθεση ε, καθώς ε, ουσιαστικά μπορούν να υπάρχουν πολλές ποικιλίε. Ε, οι νοθευτικές ουσίες ε, που επιλέγονται είναι σχετικά εύκολο να προσθεθούν και υπάρχει μεγάλη δυσκολία να τις εντοπίσουμε. Έτσι, λοιπόν, το να ελέγχουμε τα κριτήρια της σύνθεσης δεν αρκούν πάντα για να καθορίσουμε τις κατηγορίες των ζαχάρων. Θα πρέπει να έχουμε ένα καλό επίπεδο ευαισθητοποίησης και αυτό παραμένει τεχνική πρόκληση η αναλυτική μέθοδος για την ανείχνευση δεν γίνεται με μία και μόνη μέθοδο, είναι πάντοτε ένας συνδυασμός αναλύσεων. Βασικά θα πρέπει να αρχίσεις με τη μέτρηση των φυσικών και χημικών παραμέτρων όπως η υγρασία, εγωγημότητα κτλ. Κατόπιν να προσθέσεις μικροσκοπική εξέταση για να ελέγξεις τη δηλωμένη βοτανική πηγή μέσω ανάλυσης της γύρης Επιπρόσθετα θα πρέπει να καθορίσει το περιεχόμενο της ζάχαρη μέσω χρωματογραφίας για να έχουμε το προφίλ της ζάχαρης, ε, του μελιού και πρέπει αυτό να το συγκρίνεις με βάση δεδομένων που συνδέουν με τη γεωγραφική προέλευση και με το είδος των φυτών από τα οποία προέρχεται το μέλι. Επίσης, θα πρέπει να ανοιχνεύσεις την παρουσία ξένων ζαχάρων, χρησιμοποιώντας κάποιες ε, μεθόδους, ε, όπως είναι η ανάλυση αναλογίας ισοτόπου άνθρακα. Έτσι λοιπόν, ένα συνδυασμό αυτών των ε, μεθόδων μας βοηθά για να βρούμε το αν υπάρχει νοθεία στο μέλι, αλλά όλα αυτά κοστίζουν και είναι και χρονοβόρα. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα ενός... Ε, ε, έχουμε ε, μεταξύ 100 και 200 ευρώ κόστος για την ανάλυση ενός δείγματος. Λοιπόν, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα συντονισμένο σχέδιο ελέγχου που οργανώθηκε το 2015-2016. Έχει συλλέξει εμπειρία μέσω του σχεδίου δράσης ε, για το κρέας αλόγου και έτσι μπόρεσε να εντοπίσει πού έγκυτο το ζήτημα και το πού θα μπορούσαμε να ε, οργανώσουμε ένα νέο σχέδιο ελέγχου. Επιλέχθηκε το μέλη το 2014 μαζί και με κάποια ε, ψάρια. Το Μάρτιο του 2015 ε, αποφασίσαμε να συστήσουμε αυτά τα δύο σχέδια ελέγχου. Εμείς από έχουμε συμφωνήσει σε ένα εναρμονισμένο πρωτόκολλο δοκιμής και σε μια εναρμονισμένη στρατηγική δειγματοληψίας μαζί με τα κράτη-μέλη και το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο. Ο στόχος ήταν να αξιολογήσουμε την επικράτηση στην αγορά με ιού που έχουν νοθευτεί με ζάχαρα και με ιού που φέρουν λαθασμένες ετικέτες σε σχέση με τη βοτανική τους προέλευση ή και τη γεωγραφική τους προέλευση λαμβάνοντας υπόψη τα όρια των σημερινών μεθόδων για να εντοπίσουμε όλα τα είδη των ζαχάρων που χρησιμοποιούνται για νόθευση, σας ανέφερα τέσσερα βήματα στην ανάλυση. Ε, Αυτέ είναι οι μέθοδοι που υπάρχουν σήμερα ε, και το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο έχει εντεταλθεί να ερευνήσει 1.200 δείγματα μεταξύ αυτών που συλλέχθηκαν με τις εναλλακτικέ μεθόδους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε πιο αυτοματοποιημένους και αποτελεσματικούς τρόπους. Έτσι λοιπόν το σχέδιο ελέγχου έχει συλλέξει 2.300 δείγματα έχουν συλλεχθεί και από τα κράτη-μέλη και από την GRC. Αυτό χρηματοδοτήθηκε το σχέδιο 50% από την Κομισιόν ε, και από τα κράτη-μέλη. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη μελέτη, γιατί ε, δεν έχουμε βρει μια μελέτη τέτοιου μεγέθους στις διαθέσιμες δημοσιεύσεις. Είναι μια πολύ μεγάλη μελέτη που υλοποιείται, δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Πολύ συχνά ε, από άλλες μελέτες ε, είχαμε πάρα πολύ περιορισμένο σύνολο δειγμάτων σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Ήδη έχουμε προκαταρκτικά αποτελέσματα που έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα μας. Έτσι λοιπόν έχουμε 2.500 περίπου δείγματα ε, που έχουν συλλεχθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν τεθεί σε δοκιμές από τα 28 κράτη-μέλη, την Ορβηγία και την Ελβετία. Ε, τα δείγματα ελήφθησαν από την 1η Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου 2015 από εισαγωγή, παραγωγούς, ε, ε, εμπόρους, λιανικής, διανομής, από συνοριακά φυλάκια. Εμείς είδαμε ότι η απάτη κυρίως σχετιζόταν με τη δήλωση της βοτανικής προέλευσης όπου 7% θεωρείται ότι είχαν λάθος ε, ετικέτα και νόθευση με ζάχαρη 6% εντοπίστηκε στο πρώτο στάδιο της ανάλυσης. Επίσης είχαμε λιγότερο συχνή μισή μόρφωση σε σχέση με το γεωγραφική προέλευση, 2% αλλά είναι πιο δύσκολο να ερευνηθεί αυτό. Επιπρόσθετα 11% των ε, δειγμάτων που απομένουν θεωρήθηκαν ότι ήταν ύποπτα για προσθήκη ζαχάρων, αλλά με τη σημερινή μέθοδο δεν μπορούμε σίγουρα να το πιστοποιήσουμε αυτό. Το επίπεδο των υποπτών μελιών είναι πιο μεγάλο για δείγματα που ελήφθησαν σε σημεία συνοριακής διέλευσης 29% σε σχέση με άλλα δείγματα που ελήφθησαν από άλλα σημεία της διατροφικής αλυσίδας 8-10%. Έτσι λοιπόν αν θέλετε έχουμε πιο λεπτομερή αποτελέσματα ε, στην ιστοσελίδα της ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΣΑΛΤΕ σε σχέση με τις απάτες των τροφίμων. Βλέπετε ότι έχουμε υψηλά ποσοστά, μεγάλο αριθμό υπόπτων βημάτων που δεν μπορούσαμε να τα ταυτοποιήσουμε και έτσι λοιπόν δεν μπορούμε τώρα να καταλήξουμε σε ξεκάθαρα αποτελέσματα. Απλώς φυσικά ότι το επίπεδο της μη συμμόρφωσης είναι τουλάχιστον 6%. Πρέπει να ερευνήσουμε περαιτέρω και τα δείγματα και άλλα δείγματα που σέβονται τους κανόνες για να αξιολογήσουμε καλύτερα την κατάσταση. Αυτές οι πρόσθετες αξιολογήσεις και τα εργαστηριακά τεστ συνεχίζονται στο GRC. Περίπου το ίμιση από τα 200.000 δείγματα έχουν ήδη αναλυθεί και δοκιμαστεί και συνεχίσουμε τώρα την ανάλυση και θεωρούμε ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι. Η στενή συνεργασία με τα εργαστήρια στα κράτη-μέλη που έχουν εμπλακεί στο πρώτο στάδιο του σχεδίου ελέγχου έχει συσταθεί για να μας επιτρέψει την πλήρη εκμετάλλευση των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί. Η Κομισιόν θα εξετάσει την έκθεση του JRC που θα είναι διαθέσιμη μέσα τα μέσα του καλοκαιριού και σε ό,τι αφορά τα ενοποιημένα αποτελέσματα της δοκιμής, αλλά και τις συστάσεις που αφορούν την ανάπτυξη μεθόδων για τους επίσημους ελέγχους για την αυθεντικότητα του μελιού. Σε αυτή τη βάση η Κομισιόν σκοπεύει να εξετάσει το αν χρειάζεται περαιτέρω ανάληψη δράσης. Η Κομισιόν δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι το μέλι που κυκλοφορεί στην αγορά σέβεται τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρει και την κατάλληλη ετικέτα. Είναι σημαντικό αυτό για να υπάρχει ομαλή λειτουργία της αγοράς και εμπιστοσύνη στο επίπεδο των καταναλωτών. Ε, ε, μας δώσατε εκτενείς πληροφορίες. Ε, τέσσερις συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο. Η κυρία Πετήρ, Έρλ, Μπούντα, Τόρφμαν. Αλλά ένα λεπτό καθένα, παρακαλώ, μην το υπερβείτε. Κυρία Πετήρ, πρώτα. Ευχαριστώ. Οι Κροάτες μελισσοκόμοι ε, παράγουν αρκετές χιλιάδες κιλά περισσότερα από ό,τι χρειάζεται, αλλά παρόλα αυτά έχουμε μεγάλο ποσοστό που εισάγεται. 12.000 τόνους εισάγαμε είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από τρίτες χώρες στην Κροατία και μάλιστα και από την Κίνα έχουμε εισαγωγές μέλιου. Το εισαγόμενο μέλι φυσικά είναι πολύ χειρότερη ποιότητα από το ντόπιο και μάλιστα είναι και ακριβότερο ε, γιατί προβάλλεται ως ε, ιδιαίτερα ποιοτικό, κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Γι' αυτό ε, θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται να θέσει πιο αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου σε ό,τι αφορά κυρίω την επισήμανση τη χώρα προέλευση του μελιού. Το επισημάνομαι και άλλη φορά στη Γεωγραφική Επιτροπή, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ω ε, ε, τόπος προέλευση του μελιού δεν είναι αρκετό σήμα, απλώς μέλη προέλευσης, ε, ως τοποθεσία προέλευση. Γιατί ακόμη και μέλη προέλευση τρίτων χωρών τίθεται στην αγορά, στην αγορά ως μέλη Ευρωπαϊκής Ένωση. Ο κύριος Έρντο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε και κύριοι. το μισό από το μέλι που εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μισό από το μέλι το οποίο καταναλώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχεται από το εξωτερικό. Μόνο κατά το ίμιση μπορεί να πούμε ότι έχει παραγωγή ευρωπαϊκή στην καταναλωσή τη και βέβαια μεγαλώνει και το ποσοστό των απατών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει εποπτεία, είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλάβει δράση στην υπόθεση των απατών γιατί είναι απαραδεκτό να μην μπορεί να διερευνηθεί και να αποδειχθεί ποιος κάνει απάτες. Ασφάλεια στην αλυσίδα των τροφίμων δεν μπορούμε να έχουμε αν δεν μπορούμε να ελέγξουμε κάθε κομμάτι της αλυσίδας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα φαινόμενο πολύ δεδομένο και στη Ρουμάνια. Πριν από ένα μήνα περίπου έγιναν έλεγχοι ε, σε διάφορα σούπερ μάρκετ και φαίνεται ότι για το μέλια κακίας ήταν τελείως παραπλανητική η ετικέτα, γιατί το μέλι ακακίας υποτίθεται ε, περιείχε και γλυκόζη, σιρόπι γλυκόζης βιομηχανικής προέλευσης, κάτι που δημιουργεί και υγειονομικά προβλήματα. Προσοχή λοιπόν, και κινδύνου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εντατικοποιήσει τον έλεγχο και να γίνεται πιο ποιοτικό και πιο σοβαρός. Στη Ρουμανία οι μελισσοκόμοι αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες ε, το των μεγάλων ποσοτήτων νοθευμένου μελιού που κυκλοφορεί στην αγορά. Δεν έχουμε αρκετού μηχανισμού για να αναχαιτήσουμε τέτοια φαινόμενα νοθεία. Θα πρέπει να αντιδικοποιήσετε λοιπόν του ελέγχου, σα ε, παρακαλώ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Στροφάνη Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μεδιατέρος ε, που ασχολούμαστε με το θέμα αυτό. Αρκεί να κοιτάξει κανείς σε ένα σούπερ μάρκετ ποια ποσοστά και την προέλευση του ε, που πωλείται. Ε, το θέμα της κυρίας Πετήρ επίσης της σήμανσης ιδιαίτερα θέλω να επιμείνω. Πρέπει πέραν της χώρας προελεύσεως ε, που μπορεί να αναγράφεται να κοιτάξουμε τα μείγματα μελιών γιατί υπάρχει από ό,τι μαθαίνουμε δυνατότητα να απολυθεί μέλι, το οποίο είναι μείγμα από εγχώριο και μη ευρωπαϊκό. Και μάλιστα μερικές φορές το ευρωπαϊκής προελεύσεως μέλι ε, είναι σε πολύ μικρές ποσότητες τα μείγματα αυτά, έως και ομοιοπαθητικής ε, ε, ποσότητας. Μπορεί να έχουμε δηλαδή ένα κιλό ακόμη ή περισσότερο από το κινέζικο μέλι και ένα ελάχιστο ποσοστό γραμμάρια μόνο από το ευρωπαϊκό. Δεν μπορεί λοιπόν αυτό να μην καταγράφεται με ξεκάθαρους χαρακτήρες ε, πάνω στη συσκευασία για να γνωρίζει ο καταναλωτής χρειάζεται η σήμανση προλέψεως να είναι πάρα πολύ σαφής. Ευχαριστώ Σάντρα Ροντρίγκε. Ένα λεπτό κι εσείς. Ευχαριστώ. Και εγώ έχω μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί στη Γαλλικία οι μελισσοκόμοι ε, βασίζονται θορυβημένοι και προβληματίζονται με αυτή την κατάσταση των δόλων πρακτικών και της νοθείας στο μέλι. Διαρωτώνται λοιπόν οι μελισσοκόμοι πώς είναι δυνατόν να έχουμε τόσο φθηνό, με, τόσο φθηνό εισαγόμενο μέλι αν δεν κρύβεται πίσω από αυτό μια δόλια πρακτική νοθεία. Επίση, ποια είναι η θέση τη Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα τη ετικετοθεσία. γιατί ε, πολλές φορές έχουμε μέλη που δεν αναφέρει την προέλευση, τη χώρα προέλευση. Φαντάζομαι ότι ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημείωσε με προσοχή τι παρατηρήσει και τι ερωτήσει των Ευρωβουλευτών. Θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί πάνω από όλου του ελέγχου μα Φαντάζομαι θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό και θα συζητήσουμε να συμπληρώσετε τις πληροφορίες. Τώρα, αν έχετε κάποια ιδιαίτερη παρατήρηση να την κάνετε τώρα, έχετε την ευκαιρία, αλλά σας θέρμο παρακαλώ επιγραμματικά. Thank ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα απαντήσω βεβαίως ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να συζητήσουμε με βάση τα δεδομένα. Θα έχουμε τη σχετική ε, έκθεση για τα 29 άτομα ε, μπορεί να έχουμε για το 29% πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία, μπορεί να είναι και 22, μπορεί να είναι και λιγότερο ή περισσότερο. Άρα να έχουμε στοιχεία και να επανέλθουμε να δώσουμε απαντήσεις Σα ευχαριστώ. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Το φθινόπωρο. Όταν ε, δημοσιευθούν τα επόμενα αποτελέσματα των μελετών σας. Σα ευχόμαστε καλή επιτυχία στις ε, έρευνες. Οι σε μα έδωσαν ένα επιπλέον δεκάλεπτο. Κύριε Χόισλινγκ, να αρχίσουμε σήμερα την ενημέρωση και να τη συνεχίσουμε αύριο ή να την αναβάλουμε καλύτερα για αύριο. Εσείς τι προτείνετε. Με ξαφνιάζει, Πρόεδρε, το ότι το βλέπω πάλι στην ημερήσια διάταξη. Φαίνεται πως πάλι προβλέπεται κάθε φορά στην ημερήσια διάταξη. Ίσως ε, θα ήταν σκόπιμο να κάνουμε κάπως πιο δομημένα τις ε, συζητήσεις. Ε, είναι λίγοι συνάδελφοι, δεν νομίζω ότι έχει νόημα να ανοίξει η συζήτηση τώρα. Σε 30 δεύτερα βεβαίως μπορώ πολύ στο αν θέλετε να σας περιγράψω τα αποτελέσματα της τελευταίας συνάντησης του τριμερούς διαλόγου, αλλά θα χρειαστεί περισσότερη συζήτηση κάποια άλλη στιγμή. Θεωρώ ότι αύριο μπορούμε να βρούμε χρόνο, έχουμε τις ψηφοφορίες αλλά θα μπορούσαμε να βρούμε κάποιο χρόνο να ζητήσουμε τη γνώμη και του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ας το αναβάλουμε λοιπόν καλύτερα για αύριο. Γιατί το θέμα είναι πολύ σημαντικό και καλό θα είναι να είμαστε περισσότεροι στη συζήτηση. Θα ήθελα παρακαλώ να διαμηνήσετε το σχόλιο αυτό στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ίσως να ακούσουμε τώρα μια και είστε εδώ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο σχόλιο για το θέμα αυτό και ο κύριος Χόισλινγκ να μας ενημερώσει αύριο. E, e, Καλά, θα αφήσουμε καλύτερα για αύριο. Η κυρία Ράνς Καρσία. Κύριε Πρόεδρε, εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτή η συζήτηση και θα προτιμούσα να την κάνουμε τώρα. Γιατί αύριο έχω πρόβλημα με το ωράριο. Και αν το αναβάλουμε για αύριο, τουλάχιστον είναι το πρώτο σημείο μετά τις ψηφοφορίες. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσω να είμαι παρούσα. Και γι' αυτό ακριβώ έμεινε στη συνεδρίαση. Και παρόλο που έχω ένα συγγενή μου άρρωστο και μόλις μπήκε και στο νοσοκομείο, Παρ' όλα αυτά ήθελα να μείνω εδώ για να λάβω μέρος στη συζήτηση. Αν την αναβάλουμε για αύριο, σας θέλουμε παρακαλώ το πρώτο σημείο μετά τις ψηφοφορίες για να μπορέσω να πάρω και εγώ μέρος. Καλώς έτσι θα γίνει. Οπότε το πρώτο σημείο μετά τις τροπολογίες θα είναι η ενημέρωση από τον κύριο Χόισλινγκ για τους τριμερείς διαλόγους. Ωραία. Ραντεβού αύριο στις 9. Μην ξεχάσετε παρακαλώ τις κάρτες σας για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Καλό σα απόγευμα.